Okay, Αγαπητοί συνάδελφοι. Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας και να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις του Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονιστών. Όσον αφορά τις ιδέες των συντονιστών, για την επιτροπολογία. Η ρυθμιστική διαδικασία για την ασφάλεια σε αερομεταφορές πήραμε μια επίγουσα αίτηση για να υπάρξει μια ε, πρώιμη χωρίς αντίδραση απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το σύστημα για την αποφυγή των συγκρούσεων στον αέρα όπως προβλέπεται στον κανονισμό 1332 Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι μετά την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου η υπεύθυνη επιτροπή θα υποβάλει μια σύσταση όσον αφορά την ε, ε, πρώιμη χωρίς αντίθεση έγκριση. Ο πρόεδρος θα ενημερώσει την Ολομέλεια των πιο σύντομα όταν μια πολιτική ομάδα ή 40 μέλη είναι κατά μια τέτοια σύσταση. Οι συντονιστέ συμφώνησαν να προτείνουν στην Επιτροπή να αναθέσει στον πρόεδρο την ε, δυνατότητα να ισχύσει αυτή η διαδικασία για το κείμενο αυτό της Κομισιόν στα πλαίσια της ρυθμιστικής διαδικασίας με εξέταση. Επόμενο. Καθορισμός εισηγητών. Υπάρχουν ε, μια σειρά από έγγραφα εργασίας της Επιτροπής ΝΑΙΔΙΣ 2 ερμηνευτικές ε, κατευθυντήριες γραμμές για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η Επιτροπή Περιφερειών επίσης έχει κάνει μια πρόταση για την ε, εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών, ανακοίνωση για το smart και την βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν είμαστε επί της ουσίας αρμόδιοι για καμία από αυτές τις αποφάσεις. Υπάρχει επίση ε, καλύτερη διακυβέρνηση ενέργεια αγορά, η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, η Τεχνική ε, Πρόοδο και ένα κείμενο τη Επιτροπή για το EPCIP και μία ανακοίνωση από την Επιτροπή για την ε, για τις επιτροπές ε, ε, Διαχείριση της Κομισιόν. Ε, δεν προτείνουμε να ληφθεί κάποια συγκεκριμένη δράση όλες αυτές. Επόμενο θέμα. Επισκέψα αντιπροσωπείων 12-13. Γίνεται μια συζήτηση για επισκέψεις το 13 αντιπροσωπιών. Και έχουμε ακόμη κάποιο περιθώριο και για το 12. Η απόφαση των συντονιστών ήταν ότι δεν θα γίνει καμία περαιτέρω ε, επίσκεψη αντιπροσωπείας το 12 και το 13 η Επιτροπή μας θα ζητήσει έγκριση για να στείλει τέσσερις αντιπροσωπείες, έξι μελών η καθεμία. Μία στην Washington, D.C., ε, αρχές Φεβρουαρίου, μία άλλη στη βορειοδυτική Αγγλία, η περιοχή μου, που θα είναι μέλλον 15 Ιουλίου, και οι συντονιστέ κλήθηκαν να κάνουν προτάσεις για τι άλλε δύο επισκέψεις μέχρι 4 του 12. Στα διάφορα, οι πράσινοι μίλησαν για το θέμα των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Θα, θα καλέσουμε τον Επίτροπο να μας ενημερώσει για το πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επίσης, έθιξαν το θέμα της εφαρμογής του κανονισμού για τα δικαιώματα των ε, επιβατών στους σιδηροδρόμους αποφασίσαμε να κάνουμε μια επιστολή στον Επίτροπο Κάλλερ για να ρωτήσουμε πώς έχει εφαρμοστεί ο κανονισμός στα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένου του θέματος της ενιαίας παροχής εισιτηρίων και ενιαίων τιμολογιών εισιτηρίων. Υπάρχουν ερωτήσεις όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Προέδρου για τους δανειστές. Συμφωνείτε με τις αποφάσεις όπως τις παρουσίασα. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα στη μέρη διάταξη είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκθεση για την εκπαίδευση των ναυτικών. Κατέληξαν επιτυχώς οι διαδικασίες του τρομερού διαλόγου που έγιναν στις 19 ε, Ιουνίου, παρουσία του κυρίου Κουμουτσάκου που ήταν ο σκιώδης συγητής του ΕΛΚ το Κορεπερένα συμφώνησε με το συνολικό συμβιβασμό στις 27 Ιουνίου για το συνολικό πακέτο και η συμφωνία θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον Οκτώβριο. Δεν είναι απόλυτα σαφές ε, πότε θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη για να ξέρετε τι περιέχει αυτός ο συμβασμός. αφορά την εφαρμογή κατεξοδότηση πράξεων. Οι εφαρμοστικές πράξεις, η κατεξοδότηση πράξεων. οι εφαρμοστικές θα είναι για τις τεχνικές ρυθμίσεις και για την συλλογή στατιστικών στοιχείων. Οι στατιστικές που βγάζουμε από τα στοιχεία που μας ε, αποστέλλονται θα είναι δημόσιες. Όπως θα θυμάστε, το Συμβούλιο αρχικά δεν το ήθελε αυτό. Είναι σημαντικό σημείο για τη διαφάνεια και για να υπάρχει πληροφόρηση για την κατάσταση της απασχόλησης στον τομέα των, ε, της ναυτιλίας. Βεβαίως θα είναι ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία, ακόμη περισσότερο, και αναφέρεται σαφώς ότι θα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστική ανάλυση. Η θέση του Κοινοβουλίου έγινε αποδεκτή όσον αφορά τις ε, εξαιρέσεις ε, στους χρόνους ανάπαυσης και τα όρια. Και μιλάμε βεβαίως και για τη σύμβαση για τους εργαζόμενους του Ναυτιλία του 2006. Η Επιτροπή μας επίσης έκανε μια αίτηση που συμπεριλήφθηκε στην οδηγία όσον αφορά την εκπαίδευση κατά της πειρατείας, υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, ούτω ώστε να είναι ελκυστική αυτή η εργασία για τους νέους, να αποφεύγονται οι απάτες όσον αφορά τα ναυτικά δελτία και η σημασία της ασφάλειας εν πλώ, καθώς και την κατάλληλη δηλαδή επιτήρηση της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν κατέληξαν ε, οι συζητήσεις του τριμερού διαλόγου για τις οποίες και σας ενημερώνω. Ωραία. Να ψηφίσουμε τώρα. Και θα αρχίσουμε λοιπόν με τον ενιαίο ουρανό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ερώτηση για να βάλω ακουστικά. Καλημέρα σας. Απλώς να σας πω πως έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Θα μου τη φέρουν τώρα σε λιγάκι, αλλά μέχρι τώρα σας παρακαλώ πολύ ε, να μου επιτρέψετε να ψηφίζω ε, Νατάσιο χειρός. Μην ανησυχείτε, θα τους μετρήσουμε όλους και μετά θα σας προσθέτουμε και εσάς. Όταν έρθει η κάρτα, απλώς την ενημερώστε με. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, Δεν έχω κάρτα, λέει κάποιο ε, τελικά. Καλώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Σασόλη έχει το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Κάνουμε έναν έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Ο κύριος Κουμτσάκος επίσης. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ωραία. Ωραία, δεν υπάρχουν ε, σε σε, για καμία πολιτική ομάδα παραπάνω ψήφοι. Ωραία. Εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, η συγγήτρια κυρία Φώστα. Να ξεκινήσουμε. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Μαρσίνκεβιτς υπέρ. Κατά άποχες να ελέγξουμε παρακαλώ τη 13. Άρχιτη ψηφοφορία. Παρακαλώ όσοι δεν έχουν την κάρτα τους να μου πούνε πώς ψηφίζουν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Από ποιες εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Από ποιες εγκρίνεται. 19. Πώς είπατε. Α, συμβαστική 4. Συμβαστική 4. Με συγχωρείτε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 19 κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να περάσουμε στην ε, συμβαστική 6 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 Λίχτεμπεργα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 Μάισνα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία α τώρα έχετε την κάρτα σας ωραία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56. Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα από την αρχή της τροπολογίας καλεί το ΕΔΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την εξέλιξη κτλ. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετε 8, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα Μέχρι που μιλάμε για συντονισμένο τρόπο και μετά το δεύτερο τμήμα τονίζει κτλ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Μισό λεπτό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 36 ψήφισαν, 35 υπέρ, ένας κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Ευχαριστώ κυρία Φώστα. Συγχαρητήρια. Περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα ψηφοφορίας. σχέδιο γνωμοδότηση για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων πλοήγησης με δορυφόρο. Η συγκίτρια κυρία Φώστα. Έχουμε μια προφορική τροπολογία στο 1-1. Είναι η τροπολογία Λιδεράτσικ που την έχετε μπροστά σας. Έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση για την προφορική αυτή τροπολογία. Όχι. Εντάξει, θα την ψηφίσουμε λοιπόν και είναι η 34 πλέον, η οποία, στην οποία προστίθεται υπέρ κατά αποχές, άρα λοιπόν απορρίπτεται. 35, Μάρτιν Σίνκεβιτς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε Ακόμα μία προφορική τροπολογία του εισηγητή θα είναι, είναι μπροστά σας μάλλον. Έχετε αντιρρήσεις στο να την ψηφίσουμε. Ωραία, λοιπόν, την 36 είναι την προφορική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Εισηγητής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37. Ακόμα μία που, στην οποία προσθέσετε προφορική Έχουμε αντίρρηση στο να ψηφίσουμε και την προφορική τροπολογία. Όχι. 37 συν την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Μαρσίνκεβιτς πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 επιπροσθέτως υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε λοιπόν για την 40 στην οποία, την οποία θα προσθέσουμε με την ηλεκτρονική κάρτα. Ψηφίζουμε. Έχετε ψηφίσει όλοι. Ωραία λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 41 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 9 ξεκινάει η ψηφοφορία συν μία πλην μία ωραία έχετε ψηφίσει όλοι λοιπόν λίγοι απορρίπτεται άρθρο 7 προφορική του κυρίου Λιμπεράτσκι για το 43. Έχετε αντιρρήσεις στο να την ψηφίσουμε? Όχι. Ωραία λοιπόν. 43 συν την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θα ήθελα να το ε, δούμε ηλεκτρονικά. Για την 43. Έχετε ψηφίσει λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε την ε, αρχική τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι λίγη ψηφοφορία Απορρίπτεται. 46. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, υπέρ. Στη 46. Λίχτεμπεργκερ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εύα πάμε καλά. 48. Υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 48. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι, είμαστε πάλι στην πλην μία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δέκα. Εισηγητής υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 Υπέρ. Κατά,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 Έχετε ψηφίσει. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά. Υπέρ. Με συγχωρείτε, όχι ηλεκτρονικά, διανατάσσεω χειρό. Ηλεκτρονικά θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε πρώτα διανατάσσεω χειρό, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 21-22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές την 56 λοιπόν ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη εγκρίνεται η 57 καταπίπτει 58 υπέρ κατά αποχές και την 58 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 59 της κυρία Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ 23 υπέρ επαναλαμβάνω. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 24 και οι 62 είναι επανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρι... Ε, εγκρίνεται. Με 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές την 28 παρακαλώ λέει ο πρόεδρος να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται το 2 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 41 έχει εγκριθεί και η 29 έχει εγκριθεί, 30 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 με την προφορική τροπολογία έχετε καμία αντίρρηση για τη συμπερίληψη αυτής, όχι, ωραία θα ψηφίσουμε την 3 συν την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η αρχική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 η κυρία Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ την 31 ε, ξεκίνησε η ψηφοφορία λίγη απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ξεκινάει έχετε ψηφίσει όλοι λίγοι 38 υπέρ μία κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Φώστερ. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εδώ έχουμε δύο σχέδια γνωμοδότησης της κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Εύα, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το θέμα των δημοσίων ε, συμβάσεων για τις μεταφορές, ε, τα ύδατα και τις υπηρεσίες ενέργειας είναι για τις πόλεις και κομοπόλεις μας ε, ε, από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουμε σε αυτή την περίοδο. Περί τίνος πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κάνει μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του τρόπου χορήγησης των προμηθειών. Δηλαδή να υπάρξουν κάποιες διατάξεις που να τα ορίζουν. Στην πρότασή μου αναφέρομαι σε διάφορα σημεία. Πρώτον, ξέρετε ότι προτιμώ κυρίως ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, αλλά γι' αυτό ορισμένες ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να ε, καθορίζουμε αυτό που έχει έννοια να καθορίζουμε, για παράδειγμα. Όταν ε, αναθέτονται συμβόλαια αποφασιστικής σημασίας πρέπει ε, να είναι ομοιοδότης. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προκήρυξη εάν για παράδειγμα δύο ε, προσφορές είναι πάνω από 50% τότε ίσως υπάρχει πρόβλημα ενώ αλλού είναι έως 15%. Να υπάρξει ένας ε, ευρωπαϊκός ε, κανονισμός που να λέει να είναι παντού 20-25 κτλ. θα ήταν πολύ δύσκολο και σε τελευταία ανάλυση δεν θα ικανοποιούσε κανέναν. Γι' αυτό πιστεύω ότι καλύτερα αυτό το θέμα πρέπει να αριθμίζεται σε εθνικό επίπεδο. Διότι υπάρχουν διαφορετικές εθνικές παραδόσεις σε αυτό το τομέα. Σημαντικό σημείο, περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και πολλές παροιμίες γι' αυτό, ότι ο ομοιοδότης συνήθως δεν είναι η καλύτερη προσφορά. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε ε, και να προτιμήσουμε τις προσφορές που στην ουσία δίνουν καλύτερη αξία για την τιμή. Αυτό που φαίνεται φθηνότερο στην πρώτη προσφορά κατόπιν, κατά την εφαρμογή, σε δήμους ή για περιφερειακά έργα ε, προκαλούν μεγάλα μειονεκτήματα. Διότι ορισμένα θέματα αποκλείονται από την αρχική προσφορά, αλλά μετά πρέπει παρόλα αυτά να προσθεθούν. Οπότε, μακροπρόθεσμα, ανεβαίνει το ουσιαστικό κόστος. Ο μειοδότης δεν είναι πάντα ο βέλτιστος. Ο μειοδότης μπορεί να είναι καλός εάν οι συνθήκες πληρούνται. Οι συνθήκες λοιπόν που αφορούν μια δημόσια σύμβαση. Πώς πρέπει λοιπόν να είναι η προκήρυξη. Κατά τη γνώμη μου, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης πρέπει να βελτιωθεί πολύ ε, ο τρόπος προκήρυξης. Η τέχνη της προκήρυξης δεν είναι παντού επαρκώς κατακτημένη. Διαπιστώνουμε ότι δεν λαμβάνουν υπόψη θεμελιώδη θέματα σε ορισμένες προκήρυξεις. Δεν μπορούμε με κανόνες να τα επιβάλλουμε όλα αυτά, αλλά συνοδευτικά σε αυτά που θα αποφασίσουμε θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ότι ο τρόπος ε, κατάρτισης των προκηρύξεων είναι υψηλή πολιτική τέχνη. Πρέπει να φροντίσουμε να είναι γνωστοί οι κανόνες, να έχουν αποσταλεί και η ύπαρξη ή μη ύπαρξη κανόνων έχει τη σημασία της και πρέπει να είναι σαφές. Άλλο σημείο. Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να προβλέπουν συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, η κατάργηση φραγμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών. Είναι πολύ βασικό θέμα λοιπόν για μας. Όμως αν θέλουμε να είναι πολύ αυτερά τα κριτήρια, τότε υπάρχουν δυσχέρειες για να επιβάλλουμε τέτοια κριτήρια κατάργησης φραγμών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να διατεμπώνται τα κριτήρια που να ευνοούν συγκεκριμένε επιχειρήσεις. Αλλά παρόλα αυτά να υπάρχουν κριτήρια που να αφορούν τη διαδικασία παραγωγής κάποιου προϊόντος. Για παράδειγμα να αποκλείεται η παιδική εργασία, θεμητό εμπόριο και άλλα. Αλλά πάντα λαμβάνοντα υπόψη, και, αυτό, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντα πάντα υπόψη ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι θεμητά, δίκαια. Δεν είναι δυνατόν από την πίσω πόρτα, αναφέροντας ηθικά κριτήρια, να αποκλείουμε κάποιους. Για παράδειγμα, να αποκλείουμε κάποιους που δεν είναι από την περιοχή μας. Πρέπει φυσικά να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής κριτηρίων, αλλά τα κριτήρια να μην δημιουργούν διακρίσεις. Διότι αλλιώς η ανάθεση δεν θα κατέληγε. Η διαδικασία του διαγωνισμού μάλλον θα κατέληγε. Κοιτάξαμε λοιπόν πολλά θέματα, κάτι ακόμη ουσιαστικό στις υπηρεσίες μεταφορών, αλλά και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπάρχουν ήδη πολλοί αναλυτικοί κανόνες είτε είναι ο συνολικός ε, κανονισμός για τις υπηρεσίε που αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίε, είτε οι κανονισμοί για τις συγκοινωνίες, την οποία διαπραγματευόμεθα ε, για 7 χρόνια με το Συμβούλιο, με τεράστια προσπάθεια και τελικά καταλήξαμε στη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να δημιουργήσουμε διατάξεις που να είναι αντιφατικές. Γι' αυτό Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα αυτού του λεξ σπεκιάλης διότι δεν θα είχε πιστεύω έννοια ή δεν θα ήταν υπεύθυνο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβλεψε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και για τις συμβάσεις μερικά χρόνια αργότερα αυτό που αφού το αποφασίσαμε σιγά σιγά αρχίζει να εφαρμόζεται να τεθεί ένα αμφιβόλο. Πιστεύω λοιπόν ότι ένας λέξης πεκιάλης είναι σημαντικός και σωστός διότι πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Αυτά για λόγους επικουρικότητας πρέπει να πω ή γιατί επειδή νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμίσουν κάποια θέματα καλύτερα, επιμέρους. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να διαγραφούν κάποια στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν, γιατί ορισμένες ρυθμίσεις που επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα είχαν έννοια εφόσον υπάρχουν τόσο διαφορετικές παραδόσεις ανάθεσης γιατί κανέναν δεν θα εξυπηρετούσαμε. Οπότε δεν εξυπηρετούμε το στόχο μας. Έχετε τις προτάσεις μου. Παρακαλώ για τα σχόλιά σας. Έχουμε κάποιο χρόνο ακόμη. Και οι άλλες επιτροπές το συζητάνε. Πιστεύω όμως ότι ως Επιτροπή Μεταφορών πρέπει κυρίως να μας απασχολεί αυτός ο ειδικό νόμος που αποφασίσαμε για τον τομέα μας να μην υπονομευθεί εμέσως και κάποιοι συμβιβασμοί που επιτύχαμε με το Συμβούλιο να μην τηθούν και πάλι ένα αμφιβόλο. Προσβλέπω στη συζήτηση τις προτάσεις σας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει διαφορετική διαχείριση του τομέα αυτού στις διάφορες χώρες, αλλά με χαρά θα επιχειρήσω να συμπεριλάβω τις προτάσεις σας και το, από το φθινόπωρο θα έχουμε ε, κάθε δυνατότητα για διαπραγματεύσει γιατί αυτή την εβδομάδα δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ ε, από το ΕΛΚΟ Yeah. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η ανάθεση στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη της ε, οικονομίας στην Ένωση. Η οποία οικονομία στην Ένωση είναι ιδιαίτερα ε, ιδιαίτερα ε, άκαμπτη. Θα έπρεπε λοιπόν η διαδικασία ανάθεση συμβολέων και το δίκαιο ανάθεση συμβολέων να απλοποιηθεί χωρίς βεβαίως να χαθεί η σαφήνεια και η αναγκαία διαφάνεια. Η προσαρμογή του μηχανισμού ώστε να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον, να μην γίνονται ε, αποκλεισμοί, να μην μειώνεται ο ανταγωνισμός, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να έχουμε ένα σύστημα ιδιαίτερα περίπλοκο. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ λύσεις Πρώτον, πιο αποτελεσματική ανάθεση, ούτω ώστε να έχουμε τα, τα βέλτιστα αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την σχέση μεταξύ ε, τη υπηρεσίας και τιμής, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να απλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις για τις αναθέσεις. Δεύτερον, στόχος μας πρέπει να είναι ο αναθέτων να ε, προωθεί και κοινωνικούς στόχους. Για παράδειγμα, καλύτερη χρήση των πόρων, ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, καινοτομία και ή δυνατόν τις καλύτερες συνθήκες για υψηλού επίπεδου δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Και όπως και η συγγήτρια, είμαι υπέρ των ε, πρωτοβολιών που γίνεται για την απλούστευση αυτών των διατάξεων αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις για τις τροπολογίες. Για παράδειγμα, δεν λαμβάνονται υπόψη να αναφέρονται οι διαπραγματεύσεις με τους ε, εργολάβους που ε, ενδεχομένως έχουν ήδη επιλεγεί γιατί ήταν φθηνότεροι. Είναι η πέμπτη τροπολογία αυτή, ε, προσπάθεια τροπολόγηση δηλαδή, που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων. Όπου αναφερόμαστε, όπως έχουμε ήδη αναφερθεί, στα οικολογικά ε, μέσα συγκοινωνίας. Οπότε, η ίδια η διαδικασία ανάθεσης πρέπει να καθοριστεί ακριβέστερα, διότι μπορεί να γίνει και μέσω fax, μέσω ίντερνετ. Οπότε τίθεται το θέμα πότε ακριβώς θα θεωρηθεί ότι έχει συναυθεί η σύμβαση και επίσης είναι δυνατόν ε, μια, ε, ένα συμβόλιο να χωριστεί σε τμήματα που, που έχουν προτεραιότητα που δεν έχουν. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Επίσης ε, έχει διευρυνθεί ο κατάλογος και σε επιχειρήσεις που απασχολούν ανθρώπους που ζουν σε κάτω από δύσκολες συνθήκες, για παράδειγμα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν νομίζω ότι είναι σωστές αυτές οι ε, προσθήκες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λάβει πολλές ε, κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά συμβόλαια, συμβάσεις που ανατίθενται κυρίως στον τομέα των ε, υποδομών. Συνήθως λαμβάνεται υπόψη ως μοναδικό κριτήριο ομοιοδότης σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό μας οδήγησε σήμερα ορισμένες επιχειρήσεις μας να χρεοκοπούν διότι αυτή η λογική της ε, μειοδοσίας στην ουσία λειτουργήσε ισοπεδωτικά. Τραγικές επιπτώσεις για την οικονομία είχε αυτή η πρακτική. Βεβαίως η τιμή πρέπει πάντα να μας ενδιαφέρει, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής και ανάθεσης. Καλό δεν σημαίνει πάντα και φθηνό. Ευχαριστώ κυρία Μάσινα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της. Γενικά συμφωνώ. Σημαντικές οι συμβάσεις για το μέλλον της ενιαίας αγοράς και για την Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Απόλυτα σωστό. Οποτεδήποτε εκπονούμε κείμενα θα πρέπει να απλοποιούμε. Αλλά το ζήτημα είναι αυτά τα οποία αποφασίζουμε να πρέπει να μπορούν μετά να εφαρμοστούν. Ήδη αποφασίσαμε και τον Απρίλιο για την απλοποίηση. Και η ηλεκτρονική ανάθεση βεβαίως, βεβαίως θα πρέπει να το επιτρέψουμε γιατί αυτό ευνοεί και τη διαφάνεια. Θέλουμε διαφάνεια, δεν έχουμε επαρκή. Μπορούμε όντως καλύτερα να δούμε αν προσθέτει η ευρωπαϊκή αξία μία ανάθεση αυτού του τύπου. Φυσικά δεν θέλουμε να υπάρχουν διακρίσεις, όλα είναι απόλυτα σωστά, θέλουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Απόλυτα συμφωνώ με όλα αυτά. Όπου δεν συμφωνώ απόλυτα είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το κριτήριο της ε, μειοδοσίας. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη. Ποτέ δεν ήταν το μοναδικό κριτήριο. Ούτε και στο μέλλον θα είναι. Όχι, ποτέ δεν ήταν. Ποτέ. Υπάρχουν διαφορετικές βέβαια πρακτικές στην κάτω Σαξονία από όπου είμαι είδα πια τα κριτήρια όπου η ελάχιστη τιμή είναι ένα από τα κριτήρια, αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια ποιοτικά που πρέπει να τηρούνται. Γιατί λοιπόν να το καταργήσουμε εντελώ αυτό το κριτήριο. Φυσικά πρέπει να υπάρχει βιώσιμη προσφορά και να υπάρχει καλή σχέση ε, τιμής και αποτελέσματος. Είναι δύσκολο βέβαια να υπάρχουν ε, αντικειμενικά κριτήρια σε αυτούς τους τομείς. Βιωσιμότητα βεβαίως, βεβαίως βοηθάει το περιβάλλον και στην ουσία είναι και φθηνότερο για τις ε, μελλοντικέ γενιές. Γι' αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει μείγμα κριτηρίων για να πάρουμε την κατάλληλη προσφορά. Να μην αποκλείσουμε λοιπόν την τιμή. Η συγγήτρια γράφει ότι οι αναθέτοντες θα πρέπει να ξέρουν πώς να αποφασίσουν. Ε, βεβαίως, αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η επιλογή λοιπόν. απόλυτα σωστό να καταργούνται φραγμοί, να μην υπάρχουν εμπόδια, δηλαδή έχουμε όλο και ε, γυρεότερα άτομα, θα πρέπει λοιπόν να μην τους δημιουργούμε φραγμούς και εμπόδια. Φυσικά πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό. Για την επικουρικότητα. Όλοι είμαστε υπέρ της επικουρικότητας. Το ερώτημα είναι αν είναι αυτός ο σωστός τρόπος να Υπάρχει επικουρικότητα. Το δίκαιο των συμβάσεων ε, ε, προβλέπει, όπως ξέρετε, ευρωπαϊκές, δυνατότητα ευρωπαϊκής προκήρυξης. Αν είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από κάθε χώρα, τι έννοια έχει. Βεβαίω θα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται προκήρυξη πανευρωπαϊκά. Καλά, είναι κάποιε υπηρεσίε διάσωση. Ε, εντάξει, ίσω δεν θα πρέπει να γίνεται ευρωπαϊκή προκήρυξη και κάθε χώρα έχει ε, τη δική της δομή για αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά έχει έννοια να μπορούν να γίνονται ευρωπαϊκές προκήρυξεις. Για πολλά λοιπόν θέματα συμφωνώ με την εισηγήτρια, αλλά για ορισμένα έχω κάποια ερωτηματικά. Οπότε νομίζω ότι ενδεχομένως θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαριστώ όλοι ο πρόεδρος, ο κύριος Πέρκαρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επί του ουσία συμφωνώ με την εισηγήτρια. Είναι σαφές ότι ε, θεωρεί ότι δεν πρέπει όλα αποκλειστικά να αποφασίζονται ευρωπαϊκά. Υπάρχουν εθνικές παραδόσεις, οι οποίες ε, σκοπίμως εφαρμόζονται. Για το θέμα χαμηλότερη τιμή ή καλύτερη προσφορά. Χαμηλότερη προσφορά ή καλύτερη προσφορά. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι ορισμοί. Αυτό είναι το ουσιώδες. Γιατί μπορεί ο φθηνότερος να είναι και ο καλύτερος εφόσον πληρεί τα κριτήρια που είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Αλλά πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα. Οπότε εφόσον τηρούνται τα άλλα κριτήρια, είναι χαμηλή και η τιμή, Άρα έχει να κάνει με το πώς έχει καταρτιστεί η προκήρυξη, να είναι σαφής, ούτως ώστε να είναι απλούστερη η διαδικασία ανάθεσης. Να μην υπάρχει αναγκαστικά αυτή η αντίφαση καλύτερος ή φθηνότερος. Να είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιος είναι ο καλύτερος. Βεβαίως πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες Ξέρουμε όλοι ότι πολύ συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα καινοτόμε. Κάνουν θαυμάσιες προσφορές, αλλά δυστυχώς δεν είναι σε θέση όλα αυτά τα έγγραφα και τις αιτήσει και τα έντυπα να τα συμπληρώσουν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν την σύμβαση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε οι προκηρύξεις να είναι σαφείς αλλά και απλές. Ούτω ώστε οι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας να είναι σε θέση να ε, διαγωνιστούν. Βεβαίως είμαι υπέρ και την, ε, της κατάργησης οποιονδήποτε φραγμών και εμποδίων για τα άτομα με δυσχέρειες. Βεβαίως Υπάρχουν συνδρομικοί σταθμοί που δεν μπορούν να πάνε τα άτομα. Αυτά πρέπει να πάνε ε, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Γιατί δεν είναι πάντα τόσο εύκολο για αυτούς. Βεβαίω, εφόσον αναδιατυπώνουμε τα κριτήρια των προκηρύξεων, ευθύ εξ αρχή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτά, ούτω ώστε να μην έχουμε τέτοιε καταστάσει στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουμε. Και οι δύο πλευρέ. Εάν επιλύσουμε και αυτό το πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία. Συνολικά λοιπόν, Ευχαριστώ την εισηγήτρια και υποστηρίζω την έκθεση. Ο κύριος Ντεμπάκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε και εγώ να υποβάλω μερικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια για να μπορέσουν περισσότερες εταιρείες να πάρουν μέρος στις δημόσιες συμβάσεις και να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός ε, για να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα στις δημόσιες ε, συμβάσεις ό,τι αφορά τη διαδικασία. Οπότε είχα ζητήσει να υπάρξει ευελιξία και διαφάνεια και το είχα ζητήσει στο, όταν διαβάζω τώρα την εισήγηση ε, βλέπω την πρόταση η οποία πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε την πραγματική διαφάνεια και την πραγματική ευελιξία προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, για τα οικονομικά κριτήρια της μειοδοσίας πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί τα κριτήρια αυτά είναι κάτι που έχει εγκαθιδρυθεί ε, και όχι μόνο για την καλύτερη, τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και για την βιωσιμότητα ε, των σχεδίων. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το στοιχείο σε σχέση με την ανάθεση ε, νομίζω ότι υπάρχει μια ανθρώπινη διαδικασία που βασίζεται σε ορισμένα κριτήρια τα οποία είναι πολλαπλά και όταν ε, υπερισχύει ένα κριτήριο, το θεωρούμε πιο σημαντικό, νομίζω ότι επηρεάζεται όλη η διαδικασία της ανάθεσης και αυτό πρέπει να το διατυπώσουμε στην Επιτροπή για να υπάρχει μια ισοτιμία ανάμεσα στα κριτήρια. Πέρα από αυτό, σε ορισμένες από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει το θέμα της βιωσιμότητας και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν τονίζεται αρκετά το πόσο θα είναι ε, και τι σημασία θα έχουν ε, στις δημόσιες συμβάσεις. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα, εδώ γίνεται λόγος για τις παραδόσεις, τις εθνικές παραδόσεις κατά την ανάθεση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο ε, εναρμονισμένη κατάσταση στις δημόσιες συμβάσεις. Όσο πιο εναρμονισμένη γίνεται αυτό θέλουμε να πούμε. Η επικουρικότητα και οι εθνικές παραδόσεις για μένα είναι πολύ προστατευτική ηθικό κριτήριο, δηλαδή προστατεύει κανείς τις δικές του επιχειρήσεις, ε, το δικό του τόπο κτλ. Και τι θα κάνει με τις επιχειρήσεις που έρχονται εκτός χώρας να εγκατασταθούν. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε το κριτήριο της ευελιξίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δούμε στη συνέχεια ε, πώς θα φτιάξουμε τις δημόσιες συμφάσεις με νέα τεχνολογικά μέσα όπως είναι το, το fax, τα ηλεκτρονικά κτλ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που καθυστέρησα, ήμουν σε άλλη επιτροπή, αλλά θα ήθελα να πω πως η πρόταση της κυρίας να αποτελείται από πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και ξεπερνά τα όσα είναι ο περιεριστικός όρος του μειοδοτικού διαγωνισμού που νομίζω ότι στις περισσότερες αναθέσεις κρατικών προμηθειών είναι και το κριτήριο το οποίο επιβάλλεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν και ποιοτικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας και πιστεύω πως θα έπρεπαν όλα αυτά να δώσουν μια προστιθέμενη αξία που δεν θα εξαρτώνται απόλυτα από τη χαμηλή τιμή. Είχαμε και εξαιρετικά παραδείγματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός και σε σχέση με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολλές φορές είχαμε κινέζικες εταιρείες, στις οποίες ανατέθηκαν ε, κρατικές προμήθειες πολύ σημαντικές ε, σε τομείς ευαίσθητους όπως οι συγκοινωνίες και την επόμενη ημέρα αποδείχτηκε πως ήταν αρκετά καταστροφικές αυτές οι ε, αναλήψεις. Στη Μαυρετανία, για παράδειγμα, είδα ε, την κατασκευή ενός ε, ε, λιμένα που κατέστρεψε τις παραλίες στα νότια της χώρας. Αυτή λοιπόν η υπερίσχυση του κριτηρίου της, ε, του μειοδότη νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικέ συνέπειες. Βέβαια, χάρη διαφάνεια θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πληροφορημένοι, πληροφορημένοι για το ε, τι συμβαίνει σε κάθε ανάθεση. είχαμε και περιπτώσεις που χρειάστηκε να ερευνήσει η βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών παρακολουθούμε το τι συμβαίνει με τις κρατικές προμήθειες σε περίπτωση έργων υποδομών με τα τεχνικά τεύχη, με, τις, ε, ε, με τους τεχνικούς όρους. Αυτά όλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Έχουμε εντοπίσει πως η Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση χρηματοδότησης για τα μεγάλα έργα υποδομών προβλέπει τρεις τύπους επιδοτήσεις, χρηματοπιστωτικά μέσα και κρατική προμήθεια μέσω δημόσιας ανάθεσης. Για την περίπτωση αυτή πιστεύω πως αποτελεί την καλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης παρόλο που μας εξήγησαν πως ε, αρχικά δεν είχε προβλεφθεί για τις μεταφορές, ήταν περισσότερο ανάθεση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Πιστεύω όμως πως έχουμε μια ευκαιρία, την προσφέρει η κυρία Λίχτεμπεργκερ με την ε, προσπάθειά της. Θα μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να ε, μέσω αυτών των διατάξεων της κρατικές προμήθειας να δημιουργήσουμε σε, εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό γιατί σε αυτό μας ικανοποίησε πολύ η... το κείμενο της κυρίας Λίχτεμπεργκερ, δηλαδή μέσω επικουρικότητας να μην επιστρέφουμε κάποια θέματα σε εθνικό επίπεδο, αλλά να το κρατήσουμε σε ευρωπαϊκό, γιατί μιλάμε για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα τα κριτήρια θα πρέπει να έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό είναι νομίζω το βασικό το οποίο έχω να σχολιάσω. Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις. Η έκθεση της κυρίας Λίκτεμπέργα πηγαίνει προς την κατεύθυνση, να αναγκαίο πιστεύω, να θέσουμε κριτήρια στην Ευρώπη. 90% των δημοσίων ε, συμβολέων είναι στον τομέα των έργων, κυρίως έργα υποδομών. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αξιόλογα έργα που να προστάτουν αξία για τους δήμους, ε, τις, ε, τους νομούς, τα κράτη, όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η φθηνότερη προσφορά πρέπει να παίζει πολύ αποφασιστικό ρόλο, διότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον πώς θα δαπανίσουμε τις πιστώσεις μας. Αυτά που έγιναν στο παρελθόν, ότι η φθηνότερη προσφορά αυτομάτως έπαιρνε το συμβόλαιο, οδήγησε σε σοβαρά λάθη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Βεβαίως, η φθηνότερη τιμή αλλά η καλύτερη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα άλλα κριτήρια κοινωνικά, βιωσιμότητα, αναμφίβολα. Αλλά αποφασιστική σημασία έχει και η τιμή. Καμιά φορά βεβαίω γίνονται προσφορέ dumping. Όμως εξαιρούνται. Θα πρέπει να εξαιρούνται. Διότι υπάρχουν διάφορες διαδικασίες όπου η ψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή καταργούνται. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Απορρίπτονται. Και μια μέση τιμή είναι βασικό κριτήριο και πρέπει να καθορίσουμε το επίπεδο της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Κριτήρια για το ύψος χρηματοδότησης, δηλαδή άλλα κριτήρια όταν είναι κάτι κάτω από 100.000, κάτω από ένα εκατομμύριο, τι μπορεί να αποφασιστεί, δηλαδή ανάλογα με την τιμή σε τοπικό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριο Σουλιάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω την θέση του Αντί, θα ήθελα να ε, αντιδράσω σε αυτά που άκουσα σε αυτές τις σκέψεις. Ε, μία παρατήρηση έγινε, μιλήσαμε για μια γενικά αγορά υπηρεσιών, αγορά έργων, ε, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, για τις ε, για την ενέργεια και για τις μεταφορές. Και θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ελεύθερες δραστηριότητες και ότι υπάρχει μια πραγματική αγορά με ε, όλες τις πρωτοβουλίες που εκφράζονται μέσα στα πλαίσια μιας πραγματικής αγοράς. Ωστόσο υπάρχει μια άλλη οπτική μέσα στα πλαίσια αυτής της εισήγησης που θα ήθελα να τη σκεφτούμε, δηλαδή να τη σκεφτεί η εισηγήτρια. Ε, σε σχέση με αυτά που μας προτείνει. Πρόκειται για καταρχήν το να προσέξουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές. Και αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε σήμερα ε, και πάνω σε αυτό ξέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένες πλευρές του θέματος πρέπει να τις μελετήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για μια αγορά που έχει σχέση με ένα αεροδρόμιο. Πρόκειται για τη διαχείριση του αεροδρομίου, αλλά αν γίνεται ένας διαγωνισμός για ε, μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να υπάρχουν κανόνες πάρα πολύ συγκεκριμένοι που να θεσπίζουν όλες αυτές τις δραστηριότητες και αυτό είναι το καθήκον μας μέσα στα πλαίσια της ε, σημερινής συζήτησης και πρέπει να θεσπίσουμε λοιπόν αυτούς τους κανόνες. Πρέπει να δούμε λοιπόν όλες τις ε, εμπειρογνωμοσύνες για να, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα. Είχαμε κάποιες ε, εμπειρίες. Κάνανε οι Πολωνοί μία προκήρυξη για ένα αυτοκινόδρομο που έπρεπε να είναι ένα αυτοκινόδρομο που θα έπρεπε να είναι έτοιμος για το ε, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Πήραν ε, τη φθηνότερη προσφορά, πτώχευσε η εταιρεία και παραλίγο να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν τον αυτοκινητόδρομο. Άρα το φθηνότερο είναι το καλύτερο. Υπάρχει μια ε, παροιμία στα αγγλικά, η πίκρα από την ε, κακή ποιότητα κρατάει περισσότερα από τη χαρά τη φθηνή τιμή. Όπως το λέμε γερμανικά, ή, δεν είμαι αρκετά πλούσιο για να αγοράζω φθηνά. Άρα το καλύτερο δεν είναι πάντα το φθηνό. Πρέπει να παίξουν και τα άλλα κριτήρια ένα ρόλο, τα περιβαλλοντικά. Θα ήθελα να δω και τι έχω να πει ο συνάδελφος Γκρός από αυτού. Ωραία, όλο και περισσότερο φέρνουν το λόγο. Στην αρχή ήθελα να μιλήσουν δύο. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να υπογράψω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, ότι η τιμή είναι τμήμα της αποτίμησης ε, μιας προσφοράς. Να μην απορρίπτεται η φθηνότερη Δύο θέματα θέλω να αναφέρω. Πρώτον, ο νόμος που αφορά τις προκήρυξεις. Έχουμε απευθείας ανάθεση, έχουμε ε, ανταγωνιστικό διάλογο, έχουμε άλλες διαδικασίες. Όποιος θέλει λοιπόν ε, να κάνει προσφορά για σύμβαση σε άλλη χώρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Σημαντικό λοιπόν είναι να βρούμε έναν τρόπο, ένα κάποιο τρόπο, να υπάρξει μια προσπάθεια εναρμόνισης συνολικά του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι προκηρύξεις και αναθέσεις. Το δεύτερο είναι αυτός ο κρυφός προστατευτισμός που υπάρχει σε πολλές χώρες. Μπορεί να προσφέρει κανείς υπηρεσίες, αλλά πρέπει να έχει αναγνωρισμένη έδρα στη χώρα. Βεβαίω, μπορεί να έχει κανείς όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όλα τα αναγκαία διπλώματα μηχανικού, αλλά δεν ανήκει στο επιμελητήριο της χώρας αυτής. Και να ανήκει στο επιμελητήριο πρέπει να κάνει κάτι άλλο κτλ. Καταλαβαίνετε. Όσο καλή και αν αυτή η έκθεση, όσο καλό και αν φαίνεται το αποτέλεσμα, σε ορισμένε χώρε εξακολουθούν να είναι έντονε προσπάθειε για κάποιου επαγγελματικού κλάδους να προστατεύσουν τα δικά τους. Είναι πολύ σημαντικό από πλευρά εσωτερική αγορά, από πλευρά προστιθέμενη αξία να καταργηθούν αυτά. Κάτι άλλο προ άλλη κατεύθυνση. Νομίζω ότι οι συμβάσει ε, που μπορούν να δουν απευθεία τοπικά πρέπει να αυξηθούν. Δεν είναι αναγκαίο να μπορούν όλοι να, ε, συμμετάσχουν σε όλους τους διαγωνισμούς. Πολλές φορές είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό και λιγότερο αποτελεσματικό. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Λίγα σχόλια θέλω και εγώ να υποβάλω πριν να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι στις δημόσιες συμβάσεις ένα στοιχείο κλειδί είναι η διαφάνεια ε, και θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα, για παράδειγμα στην Ιαπωνία. Εμείς αγοράζουμε εδώ ιαπωνικά τρένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν επιτρέπεται να πουλήσουμε τα δικά μας τρένα στην Ιαπωνία. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ισχύει. Η Ιαπωνία θέλει ε, να ακολουθήσει αυτή την κατάσταση κατεύθυνση και να αγοράζουμε και εμείς, ε, να αγοράζουμε εμείς ιαπωνικά τρένα. Ε, τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Έχουμε Ευρωπαίους κατασκευαστές οι οποίοι παλεύουν πραγματικά ε, για να παραδώσουν τα προϊόντα την κατάλληλη στιγμή σύμφωνα με το συμβόλαιο και εμείς λέμε εντάξει θα μπορούσατε, εμείς έχουμε τα συγκεκριμένα συμβόλαια αλλά εσείς μπορείτε να έρθετε μέσα στην Ευρώπη και να κάνετε ό,τι θέλετε με τις συμβάσεις. Όχι αυτό είναι λάθος, είναι λάθος. Και θα σας πω και την αγαπημένη μου ρίση που την, ε, με όλο το σεβασμό που τρέφω για τη Γαλλία. Λέτε ε, ε για τα... Για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Γαλλία. Έχετε δει τρένα που να μην είναι γαλλικά, έχετε δει ε, ε, διάφορες μάρκες όπου να μην λέγεται το Made in France. Ας υπάρχει κάποια διαφάνεια επιτέλους. Ας συμφωνήσουμε όλοι ε, τουλάχιστον στη Γενική Αρχή ότι το φθηνότερο δεν είναι το καλύτερο. Το να προσέχουμε τη, τα, χρήματα των φορολογημένων, ναι είναι σωστό. Κάποια μειοδοσία χρειάζεται αλλά δεν πρέπει να παρεμβαίνει το κριτήριο της ποιότητας του προϊόντος. Ε, νομίζω ότι ε, εδώ είναι το bottom line το οποίο εξετάζουμε σε σχέση με αυτή τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και στη μειοδοσία. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος κάπου λοιπόν, παρακαλώ θα μας πείτε γιατί μπορούμε, πρέπει να εισάγουμε ιαπωνικά τρένα όταν εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε προϊόντα δικά μας τρένα στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ για την εισήγηση ε, και για την γνωμοδότηση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια καταρχήν πάνω στη γνωμοδότηση και μετά να σας απαντήσω στις ερωτήσεις. Θα συμφωνήσουμε πως η χαμηλότερη τιμή δεν είναι πάντα ο καταλληλότερος τρόπος για να επιλέξει κανείς μια πρόταση. Δυστυχώς στην πράξη όμως μοιάζει να είναι πολύ δύσκολο να αποφεύγεται αυτό το κριτήριο γιατί έχουμε πολλές τυποποιημένες προμήθειες οι οποίες γίνονται σε καθημερινό επίπεδο και βέβαια εδώ επιβάλλεται το, κριτήριο, το μειοδοτικό κριτήριο ε, κάτι το οποίο επιτρέπει και να αποφεύγεται το διοικητικό άχθος ε, Προσπαθήσαμε λοιπόν να προωθήσουμε και κάποια ακόμα κριτήρια και να επιτρέψουμε και αυτό της χαμηλότερης τιμής να χρησιμοποιείται και κυρίως όταν αυτό βρίσκεται και από τις, τοποθετείται και από τις αναθέτουσες αρχές του σημαντικού όρους. Ε, νομίζω ότι οι αναθέτουσες αρχές είναι και οι καταλληλότερες για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν τα θέματα αυτά. Τώρα ε, για τους διαγωνισμούς ε, τους ποιοτικούς ε, διαγωνισμούς και κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε το κριτήριο της βιωσιμότητας. Με αυτό θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Αλλά πώς να μετρηθεί αυτό, τι είναι βιώσιμο, τι δεν είναι βιώσιμο οικονομικά, ε, μήπως το βιώσιμο θα πρέπει να εξετάζει και κάποια κοινωνικά, υπερβαντολογικά ε, κριτήρια. Αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας. Οπότε ε, θα ληφθεί υπόψη, αλλά ο ορισμός αυτός εάν παραμείνει τόσο γενικόλογος ε, ενδεχομένως να αποβεί και επικίνδυνος. Η επικορικότητα, ναι για τις δημόσιες συμβάσεις κρατικές προμήθειες είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε διαφορετικά επίπεδα ε, προμηθειών, διαφορετικά διαφορετικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, θέλουμε τουλάχιστον να εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια. Γιατί εκεί έχουμε συναντήσει τα περισσότερα προβλήματα στην καθημερινότητα με την εισαγωγή ε, της απαρχής ενός ευρωπαϊκού ορισμού που θα πλαισιώνει αυτές τις έννοιες. Θέλουμε δηλαδή να ανοίξουμε περισσότερο τις ε, αρχές ε, έτσι ώστε να ε, μπορούν οι διάφορες αρχές αλλά και οι διάφορες εταιρείες να χρησιμοποιούν αυτόν τον κοινό ορισμό σε πολλά κράτη. Και αν δεν έχουμε μια κάποια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των όρων, τότε για τους οικονομικούς φορείς θα είναι πολύ δύσκολο να περνάνε από αγορά σε αγορά και να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται ε, τα θέματα αυτά. Εξού και η εναρμόνιση λοιπόν. Μία ίσονο σημασία παρατήρηση για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, γιατί έγινε κάποια ανάφορα ε, και για τις ρυθμίσεις στο χώρο των μεταφορών αναφέρεται στη γνωμοδότηση μια οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η οποία δεν έχει καμία αναφορά στους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες. Όχι, έχει μόνο την πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ των κανόνων στην σχετική οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις κρατικές προμήθειες και σε αυτήν για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να πούμε με την επιφύλαξη του. Τώρα, για τον ε, κανονισμό για τις μεταφορές έχουμε συγκεκριμένους κανόνες για συγκεκριμένα είδη μεταφορών τα οποία γίνονται ε, με συγκεκριμένο τρόπο. Η παραπομπή γίνεται, οι αναφορές υπάρχουν, το να συμπεριλάβουμε και άλλες επιφυλάξεις ή εξαιρέσεις νομίζω θα δημιουργούσε σύγχυση Επαναλαμβάνω, πολύ τεχνική αυτή η παρατήρηση και όχι πολύ σημαντική για τα τρένα από την Ιαπωνία. Είναι ένα μεγάλο θέμα και κατανοώ πως μπορεί εκ πρώτης όψεως να επηρεάσει πολύ τις αποφάσεις σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εμπορικό εργαλείο υποδιαπραγμάτευση για να δούμε πώς μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτές τις οδηγίες και οι διαπραγματεύσεις γίνονται στο επίπεδο του ΠΟΕ σήμερα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί με διαφορετική προσέγγιση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, από ότι τα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ. Δηλαδή, έχουμε ανοίξει τις δικέ μας αγορές και προσδοκούσαμε πως και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, δεν είναι το θέμα μου αυτό, σας δίνω απλώς κάποιες βασικές πληροφορίες, αλλά στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που γίνονται στον ΠΟΕ, ζητάμε μία ισότιμη μεταχείριση μεταξύ μελών του ΠΟΕ, έτσι ώστε, εάν δεν έχουν ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση αρχικά, να το απαιτούν πλέον οι διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να επιτραπεί ε, στις ευρωπαϊκές εταιρείες να έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στη σιδηροδρομική αγορά της Ιαπωνίας, όπως έχουν οι Ιάπωνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται παραλίλω παραλλήλω με την ε, τροποποίηση των οδηγιών, γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα χειριστούμε και μια διαφορετική συζήτηση στο θέμα της δικής μας ε, πρόσβασης σε άλλες αγορές. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ έχει το λόγο. κάποιες ε, απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως θα τα πούμε στις διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες. Το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε την τιμή ως κριτήριο. Να είναι σαφές αυτό. Αλλά να ισχύει το κριτήριο τιμή πάνω από οποιοδήποτε άλλο δεν είναι το σωστό κριτήριο είναι κριτήριο που προωθεί τις προσφορές dumping, που σε τελευταία ανάλυση μετά προκαλούν τεράστιο επιπλέον κόστος. Διότι μετά έχουμε πτωχεύσεις, υπεργολαβίες κτλ. που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Οι συμπληρωματικές εργολαβίες φυσικά η φθηνότερη τιμή για κάθε δήμο, για κάθε αναθέτοντα είναι ουσιώδες. Αλλά δεν θα πρέπει. Για παράδειγμα, με βάση την αρχή της ελάχιστης τιμής, να αποκλείουμε υψηλού επίπεδου προσφορές. Ή να μην μπορούμε να έχουμε ορισμένα τμήματα αυτού, του οποίου, αυτού το οποίο θέλουμε. Λοιπόν, η καλύτερη προσφορά, η οικονομικά καλύτερη προσφορά δεν είναι κατά ανάγκη φθηνότερη. Η καλύτερη είναι αυτή που έχει περισσότερη προοπτική και υπάρχουν και μερικές ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επ' αυτού. Για παράδειγμα, είναι απόλυτα δυνατόν το κριτήριο θεμητό εμπόριο να χρησιμοποιηθεί εφόσον χρησιμοποιείται χωρίς να δημιουργεί διακρίσεις. Δηλαδή δεν ευνοούμε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Εάν λοιπόν είναι σαφής η προκήρυξη, μπορούν όλες οι εταιρείε να κάνουν σωστά προσφορέ, τις προσφορές τους. Φυσικά, έχει δίκιο ο συνάδελφος Γκρός. Βεβαίως, κάποιοι δήμοι προσπαθούν με, κάποια, κάποια, με, με την εφαρμογή κάποιων κριτηρίων να ευνοήσουν κάποιες επιχειρήσεις. Δεν είναι αυτός ο δικός μου στόχος, να είναι σαφές. Αλλά τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται σε μια προκήρυξη δεν θα πρέπει να είναι κομμένα και ραμμένα για μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν θα πρέπει δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και η απλοποίηση της διαδικασίας θα βοηθήσει. Αλλά και η βιωσιμότητα θα βοηθήσει. Να συμπεριληφθούν κριτήρια βιωσιμότητας. Τι είπε η Επιτροπή τώρα. Με συγχωρείτε που θα είμαι λίγο πιο σαφής. Όταν λέτε ότι είναι δύσκολο να το καθορίσουμε, το εξαιρούμε τότε μόνο την αρχή του φθηνότερου θα συμπεριλάβουμε. Και με τρομερές αρνητικές επιπτώσεις, dumping, ε, πτωχεύσεις, που στην ουσία δεν θα είχαμε εάν είχαμε συμπεριλάβει και άλλα κριτήρια. Η προσπάθεια να καθοριστούν τα κριτήρια πρέπει να γίνει. Αλλά θα πρέπει να τα καθορίσουμε ούτως ώστε να μην δημιουργούν διακρίσεις να μην αξιοποιούνται δηλαδή για τον αποκλεισμό εκ των προτέρων κάποιων προσφορών. Γιατί το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στην Ευρώπη αυτό. Επίσης κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι σε κάποιες χώρες ε, δεν βλέπει κανείς προϊόντα από άλλες χώρες και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία. Σωστό αυτό. Πρόκειται για, κατάχρηση κριτηρίων. Δηλαδή καθορίζονται κάποια κριτήρια με τέτοιο τρόπο ή δεν ορίζονται αρκετά επαρκώς με τρόπο ώστε να αποκλείονται κάποιοι. Κάτι άλλο. Μιλήσαμε για υπεργολάβους, βεβαίως, ή για ανάθεση κατά τμήματα. Είναι πολύ δύσκολο να το ρυθμίσουμε τι κάνουμε ούτως ώστε η αλυσίδα ευθύνης ε, να μην δημιουργεί καταστάσεις όπου κάποιοι υπεργολάβοι εάν πτωχεύσει ο γενικός ε, ε, κάτοχος του έργου να έχουν δυσχέρειες. Το έχουμε το πρόβλημα αυτό και με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και εδώ η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι αντικείμενο κατάχρησης για να ευνοούνται κάποιοι που θέλουν από την αρχή να αναλάβουν το έργο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Νομική ανασφάλεια από τον τρόπο διατύπωση των κριτηρίων. Να λάβουμε υπόψη ότι αν τα εξαιρέσουμε όλα όσα δεν έχουν επαρκώς και ποσοτικά καθοριστεί ή δεν μπορούν να καθοριστούν, τότε για το 80% των συμβάσεων δεν χρειάζεται να μιλάμε για ευρωπαϊκέ προκηρύξει και για ευρωπαϊκέ ρυθμίσει. Θα είχαμε μεγάλε δυσχέρειε. Κάποια κριτήρια πρέπει να καθοριστούν επαρκώ και είμαι αισιόδοξη θα το καταφέρουμε να μην συμπεριλάβουμε άλλα κριτήρια εκτός από το φθηνότερο δεν θα ήταν σωστό εφόσον πρέπει να έχουμε μία πιο μακροπρόθεσμη δημοσιονομική προοπτική, πρέπει να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση. Χαίρομαι λοιπόν που προσβλέπω στη συζήτηση με εσά. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε ευρεία πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Οι προθεσμίες για τις ορπολογίε είναι 18 Ιουλίου. 6 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 10 Οκτωβρίου συνεχίζει τη διαδικασία και θεωρούμε πως θα περάσει από την Ολομέλεια κάποια στιγμή το Δεκέμβριο. Νομίζω πως η πρώτη προθεσμία που θα πρέπει να σημειώσει είναι η 18 Ιουλίου για τις τροπολογίες. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα 7-8 λεπτά για να έρθει ο Υπουργός. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε στις 10.30. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, τον κύριο Ευθύμιο Φλουρέντζου. Υπουργέ, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη έχουν ε, μια ιδιαίτερη επιθυμία να ακούσουν τα όσα θα τους πείτε εσείς για την Κυπριακή Προεδρία και τις προτεραιότητες της. Ξέρω πως θα γίνει και ένα άτυπο συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώς εμείς δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά ελπίζω Υπουργέ πως ε, θα καταφέρω να έρθω ε, στην διάσκεψη ε, για την αεροπορία που θα οργανώσετε τον Οκτώβριο. Πραγματικά λοιπόν θα θέλω να σας εκφράσω τη λύπη μου που δεν θα έρθω την επόμενη εβδομάδα στη Λευκοσία, αλλά ελπίζω το όμορφο νησί σας να το επισκεφτώ τον Οκτώβριο. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το θερμό καλωσόρισμα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κύριοι Αντιπροέδροι, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ που οι θεσμοί και οι αρχές της δημοκρατίας εκφράζονται κατά τρόπο υποδειγματικό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής σας τις προτεραιότητες και τις στοχεύσεις της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών και παράλληλα να ακούσω τις δικές σας θέσεις και απόψεις. Πιστεύω ακράδαντα πως μόνο μέσα από το γόνιμο διάλογο, την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μπορεί να διαμορφωθούν πολιτικές και νομοθετήματα με γνώμονα πάντοτε μια καλύτερη Ευρώπη που να ικανοποιεί τις εύλογες προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών. Έχει λεχθεί κατά κόρον ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί την ρακοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συνεπώς, ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών με σύγχρονες και ανεπτυγμένες υποδομές είναι ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των αναγκών κινητικότητας των πολιτών και συμβάλλει στην ενίσχυση της δυνατότητας για ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περαιτέρω ανάπτυξη και η σταδιακή ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων. Κατά συνέπεια αποτελεί προτεραιότητα. Αυτά τα δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαπραγματεύσεις για την διευκόλυση συνδέοντας την Ευρώπη θα αποτελέσουν προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου οι Προέδροι του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινή τους δήλωση δεσμεύτηκαν για την όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας με κοινό στόχο την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου με επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που αποτελεί σημαντική πτυχή του υποδιαμόρφωση πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Συνεπώς θα εργαστούμε με το Ευρωκοινοβούλιο κατά τρόπο επικοδομητικό για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας σε συνάρτηση πάντα με όλες τις άλλες συνιστώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου. Η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που αποτελεί τη βασική παράμετρο της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη, αναμφίβολα θα συμβάλλει τόσο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα των μεταφορών, όσο και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη βέλτιστη διασύνδεση των συστημάτων μεταφορών προκειμένου να παρέχει πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις μεταφορών τόσο για τους πολίτες όσο και για την βιομηχανία των μεταφορών. Επί της εν λόγω νομοθετικής πρότασης, το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει επιδανικής προεδρίας γενική προσέγγιση γεγονός που αποδεικνύει ότι τα κράτη-μέλη έχουν υπερβεί τα στενά εθνικά τους συμφέροντα, προβάλλοντας την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που θα πρέπει να συνθέτει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Εκφράζουμε την ετοιμότητα μας να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή σας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας. Ο ρόλος των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κατέχει περίοπτη θέση τόσο στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική μεταφορών όσο και στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Η Κυπριακή Προεδρία στα πλαίσια άτυπης συνάντησης Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου στη Λευκοσία θα επιδιώξει να αναδείξει το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην αηφόρο ανάπτυξη των μεταφορών. Μέσα από την εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη σύζευξη, διασύνδεση δύο κεντρικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ψηφιακού θέματολογίου και της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική επιδίωξη της συνάντησής μας θα είναι η υποστήριξη των δύο πιο πάνω πολιτικών διαμέσου της προώθησης, ανάπτυξης και της χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και των ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλα τα μέσα μεταφορών. Η επιτυχής προώθηση των δυο πάνω, αναμφίβολα, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολυτροπικότητας στις μεταφορές και στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για ηλεκτρονικό σχεδιασμό της μετάβασης των πολιτών από ένα προορισμό σε άλλο κατά τρόπο αποτελεσματικό. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα παρουσιαστούν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ITS World Congress, που θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία τον προσεχή Οκτώβριο. Στην συνάντηση θα παραστούν οι δύο αντιπροεύροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σιμ Γάλλας και Νέλη Κρούς, αρμόδιοι επίτροποι για τις μεταφορές και το ψηφιακό θεματολόγιο αντίστοιχα. Έχουν προσκληθεί επίσης και οι Προέδροι των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών Τραν και Ήτρε. Θεωρούμε την παρουσία του Ευρωκοινοβουλίου στην ελόγω συνάντηση επιβεβλημένη και συνεπώς ευελπιστούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, η Προεδρία θα εργαστεί για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις συσκευές ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, ταχογράφου, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της απάτης και την μείωση του διοικητικού άχθους. Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου και μέσα από τις διεργασίες με την Επιτροπή σας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο. Αναφορικά με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρημουλκουμένων τους, η οποία όπως έχω πληροφορηθεί θα εγκριθεί αυτή την εβδομάδα από το Κολέγιο Επιτρόπων και θα αποτελείται από τρεις νομοθετικές προτάσεις, σας πληροφορώ ότι η Κυπριακή Προεδρία προσδίδει μεγάλη σημασία. Στη βάση σχετικής ενημέρωσης που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εν λόγω προτάσεις θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ότι όλα τα οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας. Επί των εν λόγω προτάσεων εκτιμάται ότι θα καταθέσουμε σχετική έκθεση προόδου στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου και ενδεχομένως να επιτύχουμε γενική προσέγγιση σε μία ή δύο εκ των προτάσεων στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην οδική ασφάλεια με επίκεντρο τους τρόπους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μεταξύ των νέων. Συγκεκριμένα η Κύπρος θα φιλοξενήσει την τέταρτη Ευρωπαϊκή ημερίδα οδικής ασφάλειας στις 25 Ιουλίου το 12 η οποία με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι αφιερωμένη στους νέους. Στην εν λόγω ημερίδα θα προσκληθούν οργανώσεις νέων τόσο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης καθώς και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Στόχος είναι να καταστούν οι νέοι συνδιαμορφωτές των δράσεων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτερα στη μείωση των θυμάτων της ασφάλτου που δυστυχώς στην πλειοψηφία τους αφορούν νέους ανθρώπους. Όσον αφορά τον σιδηροδρομικό τομέα, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος στερείται σιδηροδρομικού δικτύου, η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει την εξέχουσα σημασία του συγκεκριμένου τομέα στην ανάπτυξη της πολιτικής των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί θα θέλαμε εκ μέρου του Συμβουλίου και ιδιαίτερα εκ μέρου της απερθούσας δανεικής προεδρίας να ευχαριστήσουμε το Ευρωκοινοβούλιο για την επικοδομητική του στάση και την ευελιξία που επέδειξε επί της αναδιατύπωσης της πρώτης νομοθετικής δέσμης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η Κυπριακή Προεδρία αναμένει την παρουσίαση της τέταρτης νομοθετικής δέσμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία θα θέσουμε στο Συμβούλιο για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην προώθηση της βελτίωσης των συνθήκων εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών για ένα πιο ασφαλές και υπεύθυνο εργατικό δυναμικό καθώς και σε μια κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό η Προεδρία θα δώσει έμφαση στη μεταφορά στην κοινοτική νομοθεσία των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σε σχέση με τις υποχρεώσεις κρατών λιμένα και κρατών σημαία που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας και μέσω μια νέας πρότασης για οδηγία σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας. Επί των συγκεκριμένων προτάσεων η εξέταση στο Συμβούλιο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς και ευελπιστούμε να υιοθετήσουμε γενική προσέγγιση τον Οκτώβριο. Θα εργαστούμε πολύ στενά τόσο με τη δική σας Επιτροπή όσο και με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει μερική γενική προσέγγιση ή έκθεση προόδου αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για την πολιετή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιας Ασφάλειας, ΕΜΣΑ, σχετικά με δράσεις για αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρήπαρσης, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε μια στρατηγική πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας για ένα σημαντικό θέμα που αφορά και την Επιτροπή σας. Πρόκειται για την προσπάθεια επανενεργοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα η Κύπρος ως ναυτιλιακό νησιώτικο κράτος αναγνωρίζει τη δυναμική και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αηφόρο ανάπτυξη. Η ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής προσέγγισης των θαλασσίων θεμάτων και των παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλη. Επί η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στην αηφόρο ανάπτυξη, στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην κοινωνική συνοχή των κρατών μελών, καθώς και στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αποτελεί μέρος των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Η εν λόγω προτεραιότητα θα εκδηλωθεί με την πραγματοποίηση άτυπης υπουργικής συνάντησης στη Λευκοσία στις 8 Οκτωβρίου του 2012 στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο και της Ορμόδιας Επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη. Η εν λόγω υπουργική συνάντηση στοχεύει στην επανεργοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση πολιτικής διακήρυξης, διακήρυξη της Λεμεσού, η οποία θα καταστεί ορόσημο για την διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων που θα δημιουργήσουν νέα όθηση και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτόμου αυτής πολιτικής. Πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας είναι να προσκαλέσει στην ελόγω Υπουργική Συνάντηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου οι τοποθετήσει και οι συστάσεις επί της εν πρωτοβουλίας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών η πλήρης εφαρμογή των λιγουργικών τμήματων αέριου χώρου θεωρείται βασική συνιστόσα της διαδικασίας ολοκλήρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και ως εκ τούτου αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Στο πλαίσιο αυτό η Προεδρία θα οργανώσει συνέδριο υψηλού επίπεδου στην Κύπρο, Aviation Summit, στις 11 και 12 Οκτωβρίου και θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, ώστε να συμβάλλει καταλυτικά στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης των λειτουργικών τμήματων του εναερίου χώρου, βελτιώνοντας έτσι τις επιδόσεις των αερομεταφορών στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης της αυξανόμενης αεροπορικής κίνησης. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών αερολιμένων είναι μια σημαντική πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των αερομεταφορών. Η Προεδρία θα επιδιώξει να σημειώσει πρόοδο της διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την νομοθετική δέσμη για τους αερολιμένες, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας των αερολιμένων, τη μείωση των επιπτώσεων του θορύβου γύρω από αυτούς και την καλύτερη αξιοποίηση της χωρητικότητας τους. Επιπρόσθετα, στον τομέα των αερομεταφορών η Προεδρία στη, βάση σχετικής ανακοίνωσης που αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει την υιοθέτηση συμπερασμάτων Συμβουλίου για την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επιτυχημένη ολοκλήρωση ή επίτευξη προόδου επί των πιο πάνω νομοθετικών προτάσεων. Βασική προϋπόθεση για επίτευξη του πιο πάνω στόχου είναι η αμοιβαία, εποφελής, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη-μέλη, αλλά κυρίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης και των δυσκολιών αυτού του μεγάλου εγχειρήματο θα εργαστούμε σκληρά, με σύνεση, μέτριο φροσύνη, διαφάνεια και αντικειμενικότητα για να βάλουμε και εμείς το μικρό μας λιθαράκι στην προσπάθεια που οφείλουμε όλοι να καταβάλουμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Προσβλέπω σε μια εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και είμαι στη διάθεσή σας για να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα και να επιτύχουμε από κοινού τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης και της καινοτομίας στην πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω τις προτεραιότητες και τις στοχεύσεις της Κυπριακής Προεδρίας. Ως καλός ακροατής είμαι έτοιμος να ακούσω τις δικές σας εκτιμήσεις και απόψεις και να απαντήσω στο μέτρο του δυνατού στα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Minister, thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας στο θέμα. Τώρα θα καλέσω πρώτα, θα το λόγο στους συντονιστές πρώτα και ε, διάφορους ε, ομιλητές οι οποίοι θα παρέμβουν. Ε, θα ήθελα να κρατηθούμε στα πλαίσια του χρόνου. Καταρχήν, ο κύριος Πώς. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκρόσο, πλευράς του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, για την εισαγωγή και τις εξηγήσεις σας. Φυσικά σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την εφαρμογή του προγραμματός σας. Ιδιαίτερα λόγω της γνωστής και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας των μικρών χωρών. Χρειαζόμαστε την ε, υποστήριξή σας. Μιλήσατε για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, τα FAB. Είναι σχεδόν ε, βασική ερώτηση που κάνουμε σε όλα σε όλες τις προεδρίες πώς θα προωθηθεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Βεβαίως αναφερθήκατε επίσης στο ότι τα FABs είναι ενδιαφέροντα για την ανάπτυξη της οικονομίας, για το περιβάλλον, για την ασφάλεια. Οπότε τίθεται πραγματικά το ερώτημα. Γιατί τόσο πολλές χώρες δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτά τα FAB. Τίθεται επίσης το θέμα της αξιοπιστίας μιας νομοθετικής προσπάθειας όπου τα τρία θεσμικά όργανα θέλουν να αποφασίσουν και δεν τα καταφέρνουν. Και δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που αποφασίζουν. Θα ήθελα ω Προεδρεύον του Συμβουλίου να μας πείτε και να μας πείτε και να πείτε και στους συναδέλφους σας όχι σε αυτό το θέμα. Και όχι ε, και όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για άλλα να τους πείτε ότι πρέπει να τιμούν την υπογραφή τους. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξέρετε ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2012 ήταν η προθεσμία για να εφαρμοστούν τα ΦΑΜ, Δηλαδή το Δεκέμβριο θα έπρεπε να τα έχουμε εφαρμόσει. Θα έπρεπε λοιπόν στην επόμενη συνάντηση θα περιμέναμε από εσά πληροφόρηση για το πώς έχει προχωρήσει το θέμα αυτό. Όπως είπα, είναι η περίοδος πολύ συναρπαστική μπροστά σα γιατί πολλά ενδιαφέροντα θέματα πρέπει να περάσουν σε κατάληξη. Ε, ε, έχουμε μιλήσει για του ταχογράφου. Με ενδιαφέρει αυτό που είπατε επίση και για τι θαλάσσιε μεταφορέ. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη πολιτική, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα κοινωνικά θέματα. Να αναφερθώ λοιπόν σε αυτό το τομέα. Ω κοινοβούλιο δεν μα ενδιαφέρει μόνο η τεχνική πλευρά του ταχογράφου, αλλά υπάρχουν και κοινωνικά στοιχεία. Θα θέλαμε να τα συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Για μας, το θέμα για μα δεν είναι απλώ να βελτιωθεί αύριο η κατάσταση στις οδικές μεταφορές, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται η πολιτική μεταφορών για τι οδικέ μεταφορέ με καλύτερα κοινωνικά κριτήρια. Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο η ασφάλεια σε αυτό, το καταλαβαίνω. Του επόμενου μήνε ο συνάδελφο Κοχ έχει ένα ενδιαφέρον θέμα να υποβάλει. Περιμένουμε συγκεκριμένα βήματα να σημειωθούν. Θα ήθελα, επαναλαμβάνουμε, ξέρουμε ότι πρέπει να μειωθούν οι νεκροί και τραυματίε στου δρόμου. Θέλουμε να βελτιωθεί η ασφάλεια. Θέλουμε συγκεκριμένα όμως μέτρα πιο συγκεκριμένα όχι μόνο να μιλάμε για καλή βούληση, ίσως και άλλες μέθοδοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Το πολύ σημαντικό θέμα που εδώ και μερικούς μήνες ε, μας απασχολεί είναι φυσικά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και από την άλλη πλευρά η χρηματοδότηση αυτών των δικτύων που συνδέεται και με τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές. Απλή ερώτηση. Τις κατευθυντήρες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα το προωθήσετε όπως το πρότεινε η Κομισιόν περαιτέρω και όπως το υποστηρίζει η ευρεία πλειονότητα των ε, μελών του Κοινοβουλίου μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και δεύτερον, η χρηματοδότηση αυτών των μέτρων. Και σκέφτομαι κυρίως, ε, στο, σκέφτομαι το συνδέοντα στην Ευρώπη. Είναι πολύ νέο, πολύ σημαντικό μέσο θα το προωθήσετε με τη μορφή και με τα ποσά που προτείνονται. Θα ήθελα να μας πείτε ε, ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλκατρα. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά. Από πλευρά σοσιαλιστών, Άλκατρα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική ε, αυτή η υπόθεση και όλα τα στοιχεία που αναφέρατε. Ε, πρόκειται για θέματα τα οποία θα πρέπει για πολύ καιρό να μας απασχολήσουν αλλά και που πρέπει να υπάρξουν και κάποιες εφαρμογές συγκεκριμένες ε, στην πράξη. Σκέφτομαι τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό για παράδειγμα καθώς και ε, το θέμα των FAB ε, που θα πρέπει να, από τον Δεκέμβριο και μετά να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Ξέρουμε ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ίδια πρόοδος παντού, αλλά για την αξιοπιστία του Συμβουλίου είναι θεμελιακό πραγματικά να υπάρξει δέσμευση, πραγματική δέσμευση, ούτω ώστε να υπάρξει μια μεταβίβαση αυτών των στοιχείων για τα οποία έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις, να έχουμε έναν αρμονισμένο ενιαίο ουρανό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το περιβάλλον αλλά και για τους επιβάτες. Εάν δεν μπορούμε να σεβαστούμε τις προθεσμίες μας, δηλαδή που είναι στο πέρας του έτους, ε, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν πιο περιοριστικά μέτρα. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας κύριε Υπουργέ. Σας ζητώ λοιπόν να λάβετε συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα για να γίνουν αυτές οι εφαρμογές μέσα στις προθεσμίες. Τώρα σε νομοθετικό επίπεδο έχουμε ε, σημαντικά θέματα. Ε, που θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά και βράχει πρόθεσμα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνέλθουμε. Για τον ταχογράφο, το ψηφιακό παραδείγματος χάρη, είναι ένα πρόβλημα, πρόβλημα τεχνικής φύσεως, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τις ε, ε, οδικές ε, μεταφορές. Θέλουμε να μπορούμε να ελέγχουμε κάπως καλύτερα την, τις χερσαίες μεταφορές, τις οδικές μεταφορές για να υπάρχουν όχι μόνο ε, σε κοινωνικό επίπεδο να υπάρχει ισοτιμία, αλλά να δούμε και το θέμα του ανταγωνισμού. Υπάρχουν ορισμένοι που ξεγλιστρούν μέσα από τα ανοίγματα που αφήνει ε, η νομοθεσία. Το σημαντικό θέμα είναι ε, τα δίκτυα, τα διευρωπαϊκτικά δίκτυα και η χαρτογράφησή τους. Πώς μπορούμε να σκιαγραφίσουμε μια σωστή χαρτογράφηση και τι συνθήκες θέλουμε να επιβάλλουμε στην Ευρώπη ε, και ποιο είναι το εύρος ε, της ε, ε, Ευρώπης αυτής και γι' αυτό σας θέτω το ερώτημα του προϋπολογισμού. Μιλήσατε για τα θέματα του προϋπολογισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα γιατί θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ κρίμα να προσπαθήσουμε εδώ να δημιουργήσουμε μια χαρτογράφηση των εναερίων μεταφορών πάρα πολύ εξαπλωμένη αλλά να μην έχουμε τον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πραγματοποίηση αυτής της χαρτογράφησης. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια, ένας τέτοιος προγραμματισμός, ότι υπάρχουν χρήματα, αρκετά χρήματα, για να χρηματοδοτηθεί αυτός ο μηχανισμός που είναι διασύνδεση ολόκληρης της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να επαγρυπνούμε στο Συμβούλιο, ούτως ώστε το Συμβούλιο γενικά για τις αερομεταφορές να κάνει τις σωστές προβλέψεις και εφαρμογές. Και το θέμα της, ε, του θαλάσσιου οργανισμού και των θαλάσσιων μεταφορών μετά. Είναι ένα θέμα που περατώθηκε στο Συμβούλιο και νομίζω ότι τον Δεκέμβριο θα δοθεί οριστική μορφή ε, στη διατύπωση αυτού του θέματος και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να σας δω μετά από αυτή την προθεσμία. Για την ομάδα μας αυτές είναι οι προτεραιότητες, αυτό είναι η προτεραιότητα το θέμα των θαλασσιών μεταφορών. Δύο λόγια ακόμα, αν μου το επιτρέπετε, ε, θα είμαστε πολύ ευτυχείς που συνεργαζόμαστε και τα δύο θεσμικά όργανα θα έχουν πολύ θετικές σχέσεις. Μάλιστα για του φιλελευθέρου, κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι κύριε. Ε, σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Μα αναφέρατε τι προτεραιότητέ σα. Μετά από αυτά που είπατε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη και έχω εμπιστοσύνη για την Κυπριακή Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από λίγο είχαμε πάει στην Κύπρο μια μικρή αντιπροσωπεία τη ομάδα μου. Κάναμε συζητήσει εκεί. Δυστυχώ δεν σα είδα εσά. Χαίρομαι τώρα που μπορώ να σα δω εδώ. Πολύ καλό νομίζω, όπως νομίζω όλοι μας, είναι ότι τονίζεται τη σημασία των ε, μεσοπρόθεσμων δημοσιογραφικών προοπτικών και τη σημασία του δικτύου, των διευρωπαϊκών δικτύων και της διευκόλυνσης για την Ευρώπη. Ε, σας ε, στηρίζουμε και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε όλα αυτά όχι μόνο ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών με τις κατευθυντήρες γραμμές που είπατε, με το πυρήνα και την ε, διαβρισή του, αλλά χρειαζόμαστε και τις αναγκαίες πιστώσεις. Από πλευράς μου, από την ομάδα μου, θα ήθελα οπωσδήποτε να επιμείνετε ισχυρά εάν θέλουν να κάνουν άλλοι περικοπές. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα σε σχέση με αυτό κάτι άλλο που είναι σημαντικό πολύ για μένα την επόμενη ε, χρονιά θα έχουμε την πλωτική φάση για τα ομόλογα έργο. Είναι πολύ σημαντικό από όλες τις πλευρές, από την Κομισιόν, από εμά, από το Συμβούλιο, να πιέσουμε ούτω ώστε να επιλεγούν προγράμματα που να μπορέσει να λειτουργήσουν αυτά τα ομόλογα έργου μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτω ώστε να κινητοποιήσουμε και άλλα χρήματα για να έχουμε λοιπόν κατόπιν μετά περισσότερα για τι υποδομέ στο μεσοπρόθεσμο. Αναφερθήκατε στη καινοτομία. Βεβαίω, σε όλου του τομεί χρειάζεται, άρα και στι μεταφορέ. Βεβαίω, ευφυεί συστήματα μεταφορών μπορούν να φέρουν περισσότερη ασφάλεια στου δρόμου και να μειώσουν και την επιβάρηση του περιβάλλοντο, αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Ισχύει αυτό. Βεβαίω, ψηφιακό ταχογράφο. Βεβαίω, βελτιώνει, φέρνει αναγκαίε αλλαγέ στα φορτηγά. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει, θα διευκολυνθούν με την εισαγωγή αυτών των μέτρων, αλλά θα δούμε ότι στι διαπραγματεύσει οι μειώσει των βαρών θα παίξουν επίση ρόλο και δεν υπάρχουν αρκετέ ε, δυνατότητε διεύρυνση σε κράτη-μέλη όπου κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίε αυτόνομοι δεν χρειάζονται όλοι οι Αυτά ήθελα να πω για αυτό το θέμα θα επανέλθω. Ενιαίο Ευρωπαϊκό ουρανό, συμφωνώ όπω και οι συνάδελφοι, τον χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε. Δεν θα είναι έτοιμο τέλο του χρόνου, το ξέρουμε. Σα υπόσχομαι, γιατί ξέρω, ότι η Γερμανία και η Γαλλία ε, βεβαίω έχουν τα κεντρικά φαμπ και είναι σαν δύο κόκορε που είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Και πρέπει κάθε φορά να θυμίζω στη γερμανική κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίε παραχωρήσει γιατί αν αποτύχουν σε αυτό το τομέα αν έχουμε υπογραφές αλλά καμία εφαρμογή, είναι απόδειξη αποτυχίας. Κακό για το περιβάλλον, κακό για τα χρήματά μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τελευταίο. Σημαντικό για μένα, οι θαλάσσιες μεταφορές. Μιλήσατε για τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα των ναυτικών, γιατί μας λείπουν νέοι ναυτικοί. Μιλήσατε για το EMSA, Είπατε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τις νέες μορφές μόλις. Σας υποστηρίζει το Κοινοβούλιο. Και τελευταίο. Χαιρετίζω το ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία, διότι ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ε, ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική. Ήμουν εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον μας και πολλοί το υποτιμούν. Διότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε καλύτερα το περιβάλλον για τι μελλοντικέ γενιέ μέσω καλύτερη πολιτική στον τομέα αυτό. Και χαίρομαι που θα το προωθήσετε το θέμα αυτό από πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα σα υποστηρίξουμε πλήρω. Ευχαριστώ. Κράμαρ, 4 λεπτά για του πράσινου. Ευχαριστώ για την παρουσίαση από πλευρά τη ομάδα μα. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία για την πρώτη Προεδρία του Συμβουλίου. Πάντα είναι εξαιρετική η κατάσταση αυτή. Ε, χαίρομαι και ελπίζω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Αναφέρθηκαν διάφορα σημεία, διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε ευρωπαϊκό συνδρομικό χώρο εδώ και 30-40 χρόνια στην Ένωση. Αλλά αν ε, εξετάσουμε πώ έχει την κατάσταση, είναι όλο μπαλώματα εκεί που είναι τα σύνορα. Η ευρωπαϊκή προστέμενη αξία δεν έχει επιτευχθεί. Γι' αυτό η ερώτημα, ερώτημά μου, θα προσπαθήσετε επιπλέον τα μεγάλα προγράμματα χρηματοδότηση στον τομέα αυτό τα προγράμματα τα διαμεθοριακά να έχουν την αναγκαία προτεραιότητα που χρειάζεται, ούτως ώστε η Ευρώπη και σε αυτό το τομέα να συνεργαστεί περισσότερο. Για παράδειγμα, ανάμεσα στο Βερολίνο και το Στετίν λείπουν 35 χιλιόμετρα ηλεκτροδότηση. Δεν έχουμε λεφτά, αλλά για δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια μπορούμε να δώσουμε επιδοτήσει. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Διαμεθοριακά προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτηθούν περισσότερο, να συγχρηματοδοτηθούν. Δεύτερον, Μιλήσατε για την ασφάλεια των νέων, για τα θύματα των ε, ατυχημάτων. Έχουμε την έκθεση Κόχ στο Κοινοβούλιο εγκρίνει πριν από λίγο για την ασφάλεια στους δρόμους μας. Το Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τόνισε ότι στις κατοικημένες περιοχές πρέπει να εισαχθεί όριο 30 χιλιόμετρων. Ξέρουμε ότι ε, όταν είναι 30 χιλιόμετρα το όριο, ε, θανατηφόρα ατύχημα 5% πιθανότητα, 50-81% πιθανότητα. Συμφωνείτε με αυτό θα πείσετε και το Συμβούλιο, ούτω ώστε να εισαχθεί όριο 30, να είναι στι κατοικημένε περιοχέ αυτό το όριο και βέβαια τα ίδια, ε, οι ίδιε οι πόλεις μπορούν να αποφασίσουν πού μπορεί να υπάρχει περισσότερη ταχύτητα. Το πακέτο για του σειροδρόμους, βεβαίω, 7 χρόνια είμαι στο Κοινοβούλιο, η Κομισιόν είπε ότι μέχρι τέλο του χρόνου θα υποβάλει την έκθεση. Με σκεπτικισμό το αντιμετωπίζω. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα δεν θα συζητηθεί, αλλά φυσικά με χαρά, επειδή είμαι αισιόδοξο, θα ήλπιζα να σα απασχολήσει. Θαλάσσιε μεταφορέ, μου άρεσαν αυτά που άκουσα. Συνθήκε εργασία των ναυτικών, βεβαίω, σημαντικό. Αρμοδιότητα, οι ευθύνε των κρατών σημαία, πολύ σημαντικό. Τονίσατε την ασφάλεια στι ε, θάλασσε. Αυτό που μου άρεσε ήταν αυτό που είπατε για τι εκπομπέ. Οι θαλάσσιε μεταφορέ είναι φιλικέ προ το περιβάλλον. Μόνο όμω αν οι εκπομπέ είναι χαμηλέ. Και ξέρετε το θέμα αυτό στην Κύπρο. Ξέρετε πόσο τα μεγάλα καράβια που ε, περνάνε γύρω από, τις, ε, από τα λιμάνια σας, γύρω από την χώρα σας, δημιουργούν πολλή μόνηση. Πρέπει λοιπόν να τεθούν όρια στις εκπομπές και στις απορρίψεις. Εναέριες ε, συγκοινωνίες, αεροπορικές συγκοινωνίες. Είπατε αυξάνεται ο όγκος, αλλά αυτό δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνουμε εμείς. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δίνουν 30 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, διότι η κυροζήνη δεν πληρώνει ΦΠΑ. Αυξάνουν λοιπόν όλα. Τα κράτη-μέλη μετά πρέπει να ε, μεγαλώσουν τα αεροδρόμια, να επεκτείνουν τα αεροδρόμια. Αν είχαμε σωστή εφαρμογή τη πολιτική ανταγωνισμού, θα ήταν, ανταγωνισμού, θα ήταν αλλιώ η κατάσταση. Θα φροντίσετε να υπάρχουν σωστέ τιμέ. Θα φροντίσετε να σταματήσουν οι ανισοτιμίε του πλαισίου για τι αεροπορικέ μεταφορέ. Θα λύναμε έτσι πολλά προβλήματα και περιβαλλοντικά. Ή θεωρείτε ότι α συνεχιστεί όπω είναι η κατάσταση, συνεχιστούν οι επιδοτήσει, γιατί ίσω ε, ω νησί και εσεί επωφελείστε από τι φθηνέ ε, πτήσει. Αλλά κατά τη γνώμη συνολικά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό στην Ευρώπη. Τέλο, σα εύχομαι κάθε επιτυχία στην πρώτη σα Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Φώστερ, από τους συντονιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε ανάμεσά μας ε, και ε, αναλάβατε αυτή την πρώτη προεδρία σας. Ε, θα ήθελα να συζητήσω για ορισμένες παρατηρήσεις που μας υποβάλλατε. Νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά περιχαράξατε όλους τους τομείς των μεταφορών και μας δείξατε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, ε, κλειδιά ε, και εγώ προέρχομαι από ένα νησί και εσείς είστε από νησιωτική περιοχή, ίσως το δικό μου νησί να είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε βιομηχανία και τουρισμού και βιομηχανία και είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο νησιωτικός χαρακτήρας. Ε, έχουμε ορισμένες ε, προτεραιότητες. Υπάρχει αυτό το μικρό συνέδριο για τις ε, ευφυείς μεταφορές το οποίο προετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Προεδρία και πιστεύω ότι αυτό είναι καταρχήν θετικό. Ε, νομίζω ότι ήδη έχετε ε, προχωρήσει πάρα με πολύ ταχύ βήμα. Η Προεδρία σας παίρνει θέση στον αγώνα ε, και θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω τα σχόλια που μας υποβάλλετε. Έχω μια μικρή επιφύλαξη μόνο για το θέμα της απασχόλησης. Είχαμε ακούσει για το θέμα της ανεργίας γιατί το θέμα της απώλειας θέσεων εργασίας και Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργασία θα δούλευαν σε οποιαδήποτε βιομηχανία και στις θαλάσσιες μεταφορές είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει ίσως να αναλάβετε κάποιες ευθύνες. Ε, δεν θέλουμε να χάσουμε τη ναυτιλία λόγω σημεών από το ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου έρχονται όλο εργαζόμενοι από τρίτες χώρες όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ε, και αυτό χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή και εγώ ως ε, θαλάσσια, ως προερχόμενη από θαλάσσια χώρα και ελπίζω ότι θα γίνουν ε, συζητήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στην Κύπρο όταν θα γίνει το συνέδριο γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές και όπου θα πάρουμε πολλές πληροφορίες. Ανησυχώ ε, για την υπάρχουσα συμφωνία industry είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε. Υπάρχουν τεχνολογικά προβλήματα και υπάρχει ένα θέμα με την Βόρεια Ευρώπη, τις σκανδιναβικές χώρες και πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο έχουν φτάσει μέχρι στιγμής. Τώρα σε σχέση με την αεροπορία, με τις αερομεταφορές υπάρχει το πακέτο των αερογραμμών και θέλουμε να υπάρξει αν είναι δυνατόν κάποια αναθεώρηση των χρονοθυρίδων, ε, του πακέτου των χρονοθυρίδων και η Κατά τη δική μας άποψη δεν χρειαζόταν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, χρειαζόταν μια διαφάνεια σε ορισμένους τομείς, αλλά δεν ξεχνάμε ότι συνολικά όλοι είμαστε ε, ε καθολικοί εταίροι και ε, ε, έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο ολόκληρο. Το θέμα του Ευρωπαϊκού Ουρανού, κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί είχαμε μια ψηφοφορία και είδαμε ότι μέσα στην Επιτροπή μας θα θέλαμε πραγματικά να ξεκινήσει το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ε, ουρανού και ε, πιστεύουμε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην Ευρώπη οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, η Σκανδιναβή για παράδειγμα, πολλές βόρειες χώρες, όλοι έχουν αναλάβει υποχρεώσεις σε σχέση με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ορανό και ότι το θέμα πιστεύουμε δεν είναι μόνο για τα FABs, αλλά είναι το θέμα όλης της τεχνολογίας, της τεχνολογικής στήριξης, το θέμα των επιχειρήσεων, το θέμα των θέσεων εργασίας. Θα μπορούσαμε να πουλήσουμε τεχνολογία παραδείγματος χάρη και μιλάμε για καθολικό ανταγωνισμό και για το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής σε τελική φάση. Αυτό είναι ένα τεράστιο πακέτο πραγματικά και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητηθεί στην συνάντηση κορυφής του Οκτωβρίου ε, και προσωπικά ενδιαφέρομαι γι' αυτό το θέμα. Ε, επίσης ε, το θέμα των υπηρεσιών που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες ήταν μια έκθεση η οποία σήμερα το πρωί πέρασε από την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλα αυτά κύριε Υπουργέ και ελπίζω να έχετε κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τα θέματα που υποστηρίζετε. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα έξι μέλη που θέλουν να λάβουν το λόγο. Δύο λεπτά για τον καθένα. Θα είμαι πολύ αυστηρός. Έχουμε 15 λεπτά στο τέλος για τον Υπουργό, ο οποίος θα δώσει απαντήσεις. Αρχίζω με τον κύριο Κόπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τις ε, προτάσεις που πάνε μακριά. Νομίζω ότι τόσο σαφώς όπως το αναφέρατε εσείς ως προτεραιότητα το θέμα των αντικών μεταφορών δεν το έχω ακούσει από καμία Προεδρία προηγουμένως. Ε, μία ολόκληρη γκάμα από συγκεκριμένα μέτρα. Πέρυσι την έκθεσή μου ε, προτείναμε, ελπίζω ε, και με, περιμένω με αγωνία ποια θέματα ε, θα ε, προωθήσετε. Σημαντικό είναι αυτό που είπατε ότι θέλετε να ε, εμπλακούν οι νέοι που ακριβώς είναι θέματα. Χαίρομαι πολύ, θύματα, συγγνώμη. Χαίρομαι πολύ που αναφερθήκατε στον ταχογράφο. Φυσικά ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν τα ατυχήματα, θα υπάρχουν ατυχήματα. Ο χρόνος μέχρι να φτάσει η πρώτη βοήθεια είναι πολύ σημαντική. Είχαμε μια έκθεση πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε εσείς, εφόσον είσαστε υπεύθυνο και για τηλεπικοινωνίες και για ε, τις μεταφορές, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη που έχουν τι υπηρεσίε διάσωση και οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων και οι κατασκευαστέ του εξοπλισμού, όλοι αυτέ συνεργαστούν. Παρακαλώ, βοηθήστε μα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητηθεί το θέμα του ε, ταχογράφου του ψηφιακού που είναι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Αύριο το πρωί υπάρχει μία συνάντηση με την Κυπριακή Προεδρία και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε προβλέψει για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κουμουτσάκος. Και καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση ε, για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Μια γενική παρατήρηση. Καλωσορίζω το γεγονό ότι το πρόγραμμα που μα παρουσιάσατε διαπνέεται από την αρχή ω το τέλο του από την ευρωπαϊκή αντίληψη, από την αντίληψη τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και όχι από στενά, ε, από στενά εθνικέ προτεραιότητε και στοχεύσει. Αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για μια επιτυχημένη Προεδρία, ε, κύριε Υπουργέ. Ε, το ίδιο, η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, που είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, στο οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι εισηγητής. Ε, και θα ήθελα εδώ ε, να σας πω ότι οι κατευθυντήρες γραμμές είναι άμεσα συναρτημένες με την διευκόλυνση για την συνδέοντα στην Ευρώπη, δηλαδή με τα χρήματα που προβλέπονται σε αυτό το νέο εργαλείο, αλλά αυτό είναι συνδεδεμένο με την συζήτηση για τον προπολογισμό για τα Multiannual Financial Framework. Εκεί η Προεδρία και οι, οι συνάδελφοί σας στην Κυπριακή Κυβέρνηση που θα ασχοληθούν με αυτό το πακέτο παρακαλώ πολύ να δείξουν μεγάλη προσοχή, να ενισχύσουμε τον προπολογισμό και μέσα σε αυτόν τον ενισχυμένο προπολογισμό να ενισχυθεί ο ρόλος των μεταφορών. Μεγάλη σημασία εδώ έχει επίσης, το χρειαζόμαστε στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, το νέο καινοτόμο οικονομικό, έργο, ε, οικονομικό εργαλείο των ομολόγων έργου ε, πρέπει να προχωρήσουμε καλά και θετικά στην πιλωτική φάση εφαρμόζονται. Ε, τέλος για την ενιαία θαλάσσια πολιτική. Εδώ έχετε ένα μικρό λόμπι μέσα σε αυτή την επιτροπή. Αυτό το λόμπι το αποτελούν δύο πρόσωπα, η κυρία Μάισνερ που ήταν εισηγητής της Γενικής Πολιτικής και ο Μιλών ως εισηγητής του πρώτου χρηματοδοτικού κανονισμού. Αυτό το μικρό λόμπι ε, έχει πάρα πολλούς φίλους και θα σας βοηθήσουμε στην επιλογή που έχετε κάνει να προωθήσετε την ενιαία θαλάσσια πολιτική σε αυτό το σημείο και επειδή προέρχεστε από ένα θαλάσσιο κράτο, θα ήθελα να σα πω ότι υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον τη Επιτροπής αλλά και γενικά του Κοινοβουλίου που κατα... καταγράφηκε με πρόσφατο ψήφισμα που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια για την αντιμετώπιση τη ε, μάστιγας της πειρατείας. Ε, και απλώ θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό προβλέπετε μέσα στο πρόγραμμά σα. Ε, είναι μια ιστορικά και πολιτικά κορυφαία στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, επενδύστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επενδύστε στον κατεξοχήν δημοκρατικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαστε μαζί σας. Mr. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας και με πολύ χαρά θα συνεργαστούμε. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μιλήσατε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και το γεγονός πως αυτά θα αποτελέσουν μια βασική προτεραιότητα της Προεδρίας σας. Έχουμε βέβαια και το, τη συζήτηση για το πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία αξίζουν περαιτέρω ε, εξέτασης. Δηλαδή, ομόλογα έργου και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Κάποια κράτη συμφωνούν, άλλα κράτη-μέλη διαφωνούν. Κάποιοι το έχουν προωθήσει πολύ. Εσείς λοιπόν τι θεωρείτε για το ότι θα γίνει στην πιλωτική φάση που θα ξεκινήσει σε λίγο. Και επίσης για τη στεγανοποίηση των 10 δις ε, για τη διευκόλυνση το Connecting Europe επίσης και για τα προγράμματα. Εκεί και έχουμε πάλι μια διαφωνία στο Συμβούλιο για το πώς μπορούν αυτά τα ποσά να χρησιμοποιηθούν και αν πραγματικά θα βοηθούν βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών. Και τέλος, πρόσφατα ακούσαμε, είδαμε μάλλον μία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρήση που κάνουν τα Ταμεία Συνοχής για τους θαλάσσιους λιμένες και για το γεγονός πως τα κονδύλια αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντα με τον καταλληλότερο τρόπο. Ποια είναι τα διδάγματα τα οποία λάβατε εσείς από αυτή την έκθεση για τη μελλοντική χρήση των Ταμείων Συνοχής στα πλαίσια των ε, διευρωπαϊκών δικτύων, των ΤΕΝ. Για τα λιμάνια, Μία ακόμα παρατήρηση. Νομίζω πως θα, κάνουμε, θα πρέπει να κάνετε κάποια απτά συγκεκριμένα βήματα. Μιλήσατε για την ε, δήλωση της ε, ε Λεμεσού. Ε, δύο λόγια παρακαλώ για αυτήν ακόμα. Η κυρία Γιάλα και εγώ θα ήθελα να συνταχθώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την ανάληψη της Προεδρίας και να σας πω πως χαίρομαι και εγώ που ακολουθείτε αυτή την πολύ ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μέσα σε αυτό το τόσο περίπλοκο θέμα που είναι οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η κινητικότητα στην Ευρώπη για το Connecting Europe, για, αυτό, για αυτή τη διευκόλυνση, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί θα πρέπει να ακολουθηθούν παράλληλα οι διαπραγματεύσεις που θα επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη χρηματοδότηση μεν για τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα και παράλληλα να, ε, να πραγματευόμαστε και το πολιετές ε, πλαίσιο. Ξέρετε πως εκεί υπάρχουν εμπόδια, δηλαδή τα 10 δις τα 10 δις από τα ταμεία συνοχής Εκεί ακόμα έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και πώς αυτό το Connecting Europe μπορεί πραγματικά να περιχαρκωθούν αυτά τα ποσά και να αποτελέσει ένα εργαλείο το οποίο ε, θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε εκεί, να γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί, να έχουμε και καλύτερη συνοχή και δεύτερον να σας πω πως ξέρετε πως έχουμε δύο δυναμικές οι οποίες αυτές τις στιγμές μας πιέζουν. Πρώτα απ' όλα ε, το ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ ε, χρηματοδότηση γιατί θέλουμε καινούρια project κτλ. Αλλά έχουμε και τις αμφιβολίες που δημιουργούν τα μεγάλα ενεργειακά και τηλεπικοινωνικά δίκτυα όπου μας λένε πολλοί πως ναι, αλλά εδώ ενεργοποιούνται μεγάλες επιχειρήσεις, ας βρουν οι ίδιες τα λεφτά. Πώς θα καλύψουμε λοιπόν τις ε, περιοχές της Υπέθρου με αραιό τις αραιοκατοικημένες όπου δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα εγκατάσταση αυτών των δικτύων. Τι θα προβλέψουμε για αυτούς έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατόν χρηματοδότηση στη διάθεσή μας. Να σας ρωτήσω και το εξή για τις επιφυλάξεις που ε, εγγράφησαν στο Συμβούλιο για το ευρωπαϊκό πλεονέκτημα και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Θα πρέπει το ευρωπαϊκό συμφέρον να κυριαρχήσει και να αφήσουμε στις άκρες τους εθνικούς εγωισμούς. Ίσως λοιπόν χρειαζόμαστε μια νομική έκθεση η οποία θα... Ε, συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σκαριά μια νομική έκθεση που θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι για ε, αυτή την ε, προώθηση του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Μήπως μπορούμε εκεί κάπως να το αντιμετωπίσουμε. Έχετε προβλέψει να δείτε ποιος θα είναι ο ορισμός των τραυματιών έτσι ώστε όχι μόνο να αποφύγουμε τους θανάτους αλλά και τους τραυματισμούς από τα οδικά ατυχήματα. Τους ορισμούς λοιπόν έχετε σκοπό να τους δουλέψετε. But not least, Mr. Κύριος Δανέλης, τελευταίος αλλά σημαντικός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Υπουργέ, Καλώς ήρθατε ε, και από καρδιά σας ευχόμαστε όλοι, νομίζω, ε, καλή δύναμη και επιτυχία στην ε, Κυπριακή Προεδρία. Συνηθίζω να λέω ότι όποιος έχει βιώματα νησιωτικότητας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την ένταση και την αγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που κυρίως έχουν να κάνουν και κατεξοχήν μάλιστα με τις μεταφορές, κάθε είδους μεταφορές. Γι' αυτό το λόγο φάνηκε εξάλλου από την τοποθέτησή σας, ελπίζουμε πολύ ότι θα δώσετε όλες σας τις δυνάμεις προωθώντας όλες τις εκκρεμότητες τις οποίες και εσείς απαριθμίσατε και από εμά ακούτε. Ε, νομίζω ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που είναι μια εξαιρετικά φιλόδοξη στιγμή ε, για την Ένωση που όμως δεν πατάει καθόλου σταθερά ε, στη δική σας Προεδρία έχει ελπίδες να ε, αποκτήσει μια ε, υλοποιησιμότητα. Δεν θα μπω σε επιμέρους ζητήματα που αναφέρθηκαν εξάλλου. Να αναφέρω μόνο, μιας και λίγο πριν έρθετε ψηφίσαμε σχεδόν ομόφωνα την έκθεση της αδέλφου Φώστερ για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, ότι έχετε την δυνατότητα σε αυτήν την ε, Προεδρία να πείσετε και να πιέσετε τους συναδέλφους σας ότι δεν έχουν κανένα λόγο να συνεχίσουν τον κλεφτοπόλεμο σε σχέση με την υλοποίηση της ε, νομοθεσίας εξάλλου, ε, με την ίδρυση των FABs και τη λειτουργία όλων των συστημάτων, τη, τη στήριξη του ΣΕΖΑΡ, για όλους τους λόγους που όλοι λέμε, που όμως η γραφειοκρατία ή κάποια συμφέροντα, κλαδικά ή δεν ξέρω ποια, ε, κρατούν απόμακρη από την πραγματοποίηση αυτήν την ε, φιλόδοξη, αυτό φιλόδοξο προγραμματισμό. Ε, κλείνοντας, ε, σας διαβεβαιώ ότι το Ευρωκοινοβούλιο και ιδιαίτερος η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, είναι, θα είναι ένας βασικός ασύμμαχος στην προσπάθεια υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ε, ένα-δύο θέματα που δεν δημιουργούν δυσχέρειες, δεν είναι επίμαχα. Αλλά αν θα θέλατε να επιχειρήσετε να απαντήσετε μερικές από τις ερωτήσεις των συναδέλφων και τα σχόλιά τους, έχετε περίπου 15 λεπτά για να έχετε ένα μπούσουλα. Γιατί μετά πρέπει να συζητήσουμε για τον προπολογισμό μας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. κατηγοριοποίησης των ερωτημάτων που έχουν μπει να δώσουμε το συντομότερο δυνατό απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τα λειτουργικά τεμήματα του εναερίου χώρου, τα FAPS, γιατί έχω δει ότι πέραν από την διευκόλυνση της Ευρώπης τα ΦΑΠΣ είναι εκείνα τα οποία κυριαρχούν στις ερωτήσεις των περισσότερων και τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Όπως καλά γνωρίζετε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την εγκαθίδρυση των ΦΑΠΣ και αυτό είναι στις 4 του Δεκέμβρη το 12. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία μαζί με την Επιτροπή. Πρόσφατα είχαμε στην Κύπρο την επίσκεψη του συντονιστή των ΦΑΠΣ και την περασμένη εβδομάδα ήταν η επίσκεψη του κολεγίου και ήταν ένα θέμα συζήτησης μαζί με τον Επίτροπο Κάλλας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα για την λειτουργία των ΦΑΠΣ μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Ένας ακριβώς από τους λόγους που αποφασίσαμε να κυριαρχήσουν τα λειτουργικά τμήματα στο Aviation Summit το οποίο θα γίνει τον Οκτώβριο στην Κύπρο είναι η προσπάθεια την οποία θέλουμε να κάνουμε να αποτυπώσουμε την πρόοδο η οποία θα έχει επιτευχθεί μέχρι τότε και από εκεί μέσα από τη συζήτηση να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία θα έχουν καταγραφεί για να μπορέσουμε να φέρουμε όσο το δυνατό πιο κοντά την εγκατήθρηση των λειτουργικών τιμαμάτων. Θα δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια προς την Επιτροπή και στήριξη στην προσπάθεια για υλοποίηση των ΦΑΠΣ. Έχω ακούσει ε, για την πίεση την οποία θα πρέπει να ασκηθεί ούτω ώστε τα ΦΑΠΣ να εγκαθιδρυθούν στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί. Σίγουρα δεν μπορεί η Προεδρία να είναι εκείνη η οποία θα ασκήσει τις πιέσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή είναι εκείνη που θα ασκήσει τις πιέσεις. Εμείς θα συνεργαστούμε μαζί με την Επιτροπή σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μέχρι τις 4 του Δεκέμβρη την δυνατότητα τα ΦΑΠΣ να έχουν εγκαθιδρυθεί. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη σημασία την οποία έχουν. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει λεχθεί από αρκετούς είναι ότι θα πρέπει να προσδώσουμε αξία στην οδική ασφάλεια. Συμφωνούμε απόλυτα με την τοποθέτησή σας θα πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο της οδικής ασφάλειας. Γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό διοργανώνουμε την ημερίδα για την οδική ασφάλεια, ούτω ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους, αλλά και στους οργανωμένους φορείς, να δώσουν τις δικές τους απόψεις για τα θέματα ασφάλειας, για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν και για να καταστούν οι ίδιοι συνδιαμορφωτές αυτής της πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο θα εμβολιάσουμε και θα εμπλουτίσουμε την πολιτική της νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορές στην οδική ασφάλεια αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι στον τομέα της οδικής ασφάλειας η διαμόρφωση θα πρέπει να αρχίσει από την νεαρή ηλικία, για να μην πω ακόμα από την δημοτική ηλικία. Είναι εκεί που θα πρέπει να εναποθέσουμε τις ελπίδες παράλληλα φυσικά με όλα τα άλλα, τις άλλες πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να έχουμε υιοθετήσει και που αναφέρονται στις υποδομές, είτε αυτές αναφέρονται στα οδικά δίκτυα, είτε στα ευφυή e συστήματα, είτε άλλος πώς. Όμως, μέσα από την αγωγή στην εκπαίδευση θα δημιουργήσουμε την οδική συνείδηση που θα είναι το κλειδί για μείωση των οδικών δυστυχημάτων. Όπως γνωρίζετε υπάρχει από τον Μάρτιο μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο στη βάση μιας μεθοδολογίας που αναφέρεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και στο ΣΕΦ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να επιτύχουμε μια συμφωνία για να έχουμε δίκτυα για την περίοδο 14-20 που θα δημιουργούν ανάπτυξη και μια πραγματική προστιθέμενη αξία να συνδέσουμε δηλαδή σημαντικά σημεία στην Ευρώπη. Εμείς, αν και δεν έχουμε σαν Κύπρος ε, σιδηροδρόμους, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν τομείς μεταφορών οι οποίοι είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Η διασύνδεση των ευρωπαϊκών χωρών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διασυνδέει και δημιουργεί πραγματικά συνθήκες συνοχής, αλληλοκατανόησης των ευρωπαϊκών λαών που αποτελούν την ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχουν να συνεισφέρουν πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε υποδομές ανάπτυξης στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργειες. Οι μεταφορές καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ΣΕΦ και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα που οι μεταφορές διαδραματίζουν στον ευρωπαϊκό χώρο, γι' αυτό και αποκαλούνται και η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όσον αφορά τους ταχογράφους, υπάρχει το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μπροστά μας τις τρομπολογίες που ψηφίσατε. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσει στο Συμβούλιο. Μας αναμένουν βεβαίως και θα αναμένουμε και την μελέτη βιωσιμότητας, το feasibility study. Θα του δώσουμε την έμφαση που πρέπει για τους λόγους που είναι ε, εύκολα κατανοητοί και έχουν ήδη ηλεχθεί και από εσάς αλλά και από εμάς στην ομιλία μας. Περιμένουμε και θα περιμένουμε την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής μελέτης και θα υπάρξει ανάλογη συζήτηση στο Συμβούλιο. Θα είμαστε, κυρία Τικάο, στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών και την σύμβαση παροχής εργασίας στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. Προς εκείνη την κατεύθυνση θα εργαστούμε ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας, δηλαδή τον Σεπτέμβριο, να έχουμε γενική προσέγγιση για να αποτελέσει το εφαρτήριο για να προχωρήσει στην επόμενη Προεδρία προς ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εφαρμογή και πιστεύω ακράδαντα ότι οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, η δυνατότητα αναφοράς από τους ναυτικούς στο κράτος λιμένα για τα προβλήματα τα οποία πιθανόν να αντιμετωπίζουν δίνουν ένα υπόβαθρο όπου θα μπορούν νέοι ανθρώποι να ζητήσουν εργασία στην εμπορική ναυτιλία γιατί θα είναι θέσεις εργασίας καινούργιες με αξιοπρέπεια και που θα αισθάνονται ότι τα δικαιώματα τους είναι πλήρως διασφαλισμένα. Να έχετε τη βεβαιότητα ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε συνειδητά και σκληρά γιατί θεωρούμε ότι με την δημιουργία συνθήκων εργασίας απαυλύνουμε το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει την Ευρώπη ολόκληρη συνεπία της οικονομικής κρίσης την οποία έχουμε. I do hope that I have some more time, Mr. President. Four minutes. Four minutes. Thank you very much. I'll try my best. Ευχαριστώ. Τέσσερα λεπτά μου δίνετε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο. αρκετοί από εσά, μία από τις προτεραιότητες τις οποίες εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα όντας νησιώτικο κράτος ότι θα πρέπει να της δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Θεωρούμε ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και η επανεργοποίηση της θα είναι μια κινητήρια δύναμη που θα δώσει νέες διαστάσεις στην χρησιμοποίηση όλων των πολιτικών οι οποίες συνδέονται με τη θάλασσα. Είτε αυτές αναφέρονται στις θαλάσσιες μεταφορές, είτε αναφέρονται στην ενέργεια, είτε αναφέρονται στον τουρισμό, είτε αναφέρονται στην ηχθειοκαλλιέργεια, είτε αναφέρονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε πολλές άλλες πολιτικές. Θεωρούμε ότι με βάση τη δήλωση την οποία θα ανακοινώσουμε στη Λεμεσό στις 8 του Οκτωβρίου θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά κράτη με στόχο την ανάπτυξη γι' αυτό και την ονομάζουμε γαλάζια ανάπτυξη γιατί προέρχεται από τη θάλασσα και στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ούτω ώστε με σεβασμό φυσικά προς το περιβάλλον να υπάρξει εκείνη η ανάπτυξη και οι υποδομές που θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη του να ξεπεράσει η Ευρώπη που μας ενδιαφέρει την οικονομική κρίση να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ας μην ξεχνούμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε παράκτιες περιοχές. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλα τα δεδομένα τα οποία μέσα από την επανεργοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και με το βήμα που θα δοθεί στα κράτη-μέλη για να βάλουν τη δική τους συνεισφορά θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Ο κύριος Κουτσάκος έχει θέσει ένα ουσιαστικό για μας θέμα το οποίο έτυχε σαν Κύπρος να του δώσουμε πολύ ιδιαίτερη σημασία γιατί έχουμε ενσανθεί πολύ έντονα τις συνέπειες του και αναφέρομαι στην πειρατεία. Όπως ίσως καλά γνωρίζετε η Κύπρος έχει πολύ πρόσφατα υιοθετήσει νομοθεσία η οποία στόχο έχει την καταπολέμηση της πειρατείας ιδιαίτερα στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στις ε, παράκτιες περιοχές της Σομαλίας. Στόχος μας μέσα από την νομοθεσία η οποία έχει υιοθετηθεί είναι να προστατεύσουμε τις ζωές των ναυτικών που βρίσκονται πάνω στα εμπορικά πλοία, να προστατεύσουμε φυσικά τις ιδιοκτησίες των πλειοκτητών αλλά και τα φορτία. Όμως πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δίδουμε το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες πλοίων κάτω από την Κυπριακή σημαία να έχουν ένοπλη συνοδεία πάνω στα πλοία, ρυθμίζουμε το δικαίωμα αυτοάμυνας, ρυθμίζουμε ακόμα και τα δικαιώματα των ναυτικών οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα όταν σκάφος θα περάσει από επικίνδυνη ζώνη να μπορεί να κατέβει από το πλοίο. Δίνουμε συναμπός μέσα από την νομοθεσία την έγκριση για εταιρείε οι οποίες θα περάσουν από ένα κόσκινο για να μπορούν να παρέχουν αυτές τις ε, υπηρεσίες ασφάλειας και στοχεύουμε με αυτόν τον τρόπο να καταπολεμήσουμε την πειρατεία η οποία πλέον αποτελεί μία μάστιγα. Είναι το πλήγμα στην ναυτιλία τεράστιο λόγω ακριβώς της ύπαρξης της πειρατείας. Απόλυα ζώων, απόλυα φορτίων, απόλυα πλοίων. Αυτό επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο τα κυπριακά πλοία αλλά και όλα τα άλλα πλοία τα οποία περνούν στην περιοχή. Και εμείς μέσα από τα πλαίσια της, ε, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αλλά και μέσα από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων δεδομένου ότι η Κύπρος είναι στον τομέα της ναυτιλίας μια μεγάλη ναυτική δύναμη θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να δώσουμε τα φώτα στον βαθμό που εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ναι. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δανική Προεδρία για τη δουλειά την οποία έχει κάνει και την οποία μας έχει παραδώσει ιδιαίτερα στο νομοθετικό τομέα αλλά και εσάς, την Επιτροπή σας για την πρόσκλησή σας να είμαστε σήμερα εδώ και να δώσουμε σε αδρές γραμμές το πρόγραμμα εργασίας μας αλλά και τις προτεραιότητές μας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κυπριακής δημοκρατίας αυτό το εξάμεινο. Well, President office, can I thank you for your Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και για όλες τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των μελών. Θέλουμε πολύ και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, μετά από την Δανική και πριν από την Ιρλανδική. Εξ ονόματος, λοιπόν όλων των συναδέλφων βουλευτών που ήταν παρόντες σήμερα το πρωί θέλω να σας ευχαριστήσω και πραγματικά προσβλέπουμε, επαναλαμβάνω, στη συνεργασία μας για να υπάρχει μια επιτυχής Κυπριακή Προεδρία στον τομέα των συγκοινωνιών και έργων. Ευχαριστώ. October, but it's an overlap. Okay, Gizine. If you can be quick. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ επιστρέψτε στις θέσεις σας. Ωραία, Γκεζίνε. είναι προπολογισμό 2013, προτεραιότητε. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήδη μιλήσαμε για τον προπολογισμό. Θα ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν περικοπές και να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά είναι αναγκαίες και οι επενδύσεις και πρέπει ως μεταφορές να υποστηρίξουμε κάποιους, να υπερασπιστούμε κάποιους τομείς, να μην μας ε, τα πάρουν όλα. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο συνεδρίασε και η ομάδα εργασίας θα επιβεβαιωθεί η ομάδα εργασία από του προσβευτέ, δηλαδή τα αποτελέσματά τη στι 11 και στι 26 το Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα είναι καθαρά τυπική υπόθεση. 26 Ιουλίου λοιπόν είναι η προθεσμία, όπου με βάση την εμπειρία και των προηγουμένων ετών δεν θα αλλάξουν καθόλου την πρόταση του Συμβουλίου. Και όπω περιμέναμε, το Συμβούλιο πρότεινε σε διάφορα σημεία έντονε περικοπέ. Καταλαβαίνουμε βέβαια, το Συμβούλιο βεβαίω θέλει να περικόψει τα πάνε, αλλά πρέπει να περασπιστούμε τι προτεραιότητέ μα. Μίλησα και με τους Σκιώδη, ε, του έστειλα το κατάλογο για το τι πρόκειται να περικοπεί σε δύο σημεία. Θα μπορούσαμε κάτω από μέρε συνθήκε να συμφωνήσουμε με κάποιε περικοπέ, για παράδειγμα, υποστήριξη για προγράμματα κοινού ενδιαφέροντα για, τις, ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των μεταφορών, διοικητικέ και επιχειρησιακέ δαπάνε. Θέλουν να μειωθεί το ποσό εν μέρη. Δεν είναι σωστό, αλλά θα ήταν μια διαπραγματευτική θέση. Και επίση εξωτερικά μέτρα για την έρευνα. Θέλουν να μειώσουν κατά 200 εκατομμύρια τα άλλα σημεία που αναφέρονται για περικοπές θα πρέπει οπωσδήποτε μέσω τροπολογιών να τα εμποδίσουμε. Να εμποδίσουμε τις περικοπές. Είχαμε πει ότι δεν θέλαμε καμία περικοπή για τα TNT, για το Caesar, για την ασφάλεια της μεταφορές, για την έρευνα και για τα δικαιώματα των επιβατών. Βεβαίως, αυτά τα είχαμε προηγουμένως, θέλουμε να διατηρήσουμε οι γραμμές του προπολογισμού όπου προβλέπονται περικοπές από πλευρά του Συμβουλίου δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές από εμά. Θα υποβάλουμε τροπολογίε για να επανέλθουμε ε, στα ποσά της Κομισιόν. Αυτά είχαμε υποστηρίξει τότε. Αυτά λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε και τώρα. Έτσι έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, για τους διάφορους οργανισμούς, το Συμβούλιο ήθελε να κάνει περικοπές αλλά καταφέραμε να επανέλθουμε στα αρχικά ποσά. Είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό. Η MSA τώρα μόλις ανέλαβε ε, νέα καθήκοντα, το είπε και ο Κύπριος ε, υπουργό. Οπότε χρειαζόμαστε και τις ε, χρηματοδοτήσεις, όπως ακριβώς τις πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τους επιβάτες. Η Επιτροπή στη συνάντηση μας είπε ότι θα μας στηρίξει να παραμείνουν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Οπότε λοιπόν θα υποβάλουμε τροπολογίες στα σημεία αυτά που μόλις ε, ανέφερα, να μην γίνουν εδώ περικοπές, να επανέλθουμε στα αρχικά ποσά και από την άλλη πλευρά για τα πιλωτικά προγράμματα ακούσαμε τώρα κάτι το κάπως ε, αναπάντεχο έγινε μια πρώτη αποτίμηση των προτινομένων προγραμμάτων από τις διάφορες επιτροπές και όπως ξέρετε, σύμφωνα και με την άποψη των ε, συντονιστών είχαμε προτείνει τρία συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία έπρεπε να συνεχιστούν από τον προηγούμενο χρόνο. Προγράμματα που ήδη λοιπόν λειτουργούσαν. Δύο αφορούσαν τον τουρισμό. Το πρώτο τον τουρισμό με μια πολιτιστική και βιομηχανική πλευρά και ο δεύτερος τουρισμός για όλους, πρόσβαση για όλους και το τρίτο ήταν το ενιαίο σύστημα εισιτηρίων Ε, αλλά μας εκπλήσει το ότι η αποτίμηση των προγραμμάτων που έγινε από την Επιτροπή πήγε καλά για τα δύο πρώτα προγράμματα, αλλά για την, ε, τα, ε, πήρε το βαθμό α, δηλαδή τον πρώτο βαθμό, τον καλύτερο βαθμό, αλλά το τρίτο για το ενιαίο σύστημα ε, έκδοση εισιτηρίων πήρε βαθμό Σ, αφού είχε εγκριθεί και από πέρυσι και είχε θεωρηθεί πολύ σημαντικό. Η επιμήκυνσή του λοιπόν τίθεται εν κινδύνο. Πέρυσι η Επιτροπή Προπολογισμών είχε μόνο εγκρίνει προγράμματα που είχαν πάρει Α, 10 με τόνο. Άρα τα δύο προγράμματα του τουρισμού ε, υπάρχει περίπτωση να εγκριθούν. Άρα δεν είναι καλέ οι προοπτικέ για τα εισιτήρια. Πρέπει όμω να υποβάλουμε πρόταση και γι' αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Ίσως να μην έγινε αντιληπτή η σημασία του. Είχα προτείνει και ένα άλλο πρόγραμμα εγώ ίδια. Προπαρασκευαστικές ενέργειες. LNG για την εισαγωγή του LNG. Αυτό πήρε β βαθμό. Καλύτερα λοιπόν από τα εισιτήρια. Αλλά επειδή δεν είχα την υποστήριξη των συντονιστών για το πρόγραμμα αυτό, είχαμε περιοριστεί στα τρία που πρόκειται να συνεχιστούν. Οπότε υπέβαλα αυτή την τέταρτη πρόταση για το όνομά μου, αλλά έκανε ένα τυπικό λάθος. Ε, ε δεν διευκρίνησα ότι είναι δική μου πρόταση και όχι πρόταση των ε, συντονιστών. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Ε, θα εξετάσω τώρα εάν θα συνεχίσω, θα εμείνω σε αυτή μου την πρόταση ως προσωπική πρόταση, γιατί ε, από το βαθμό που πήρε δεν πάνε τόσο άσχημα τα πράγματα για αυτήν. Αλλά το πρόβλημα αφορά την, το ενιαίο σύστημα εκδοση εισιτηρίων. Αυτό κινδυνεύει. Αυτά προς το παρόν Αναμένω τις αντιδράσεις, αντιρρήσεις σας, σχόλια των σκιωδών ή και άλλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρίκε για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ για αυτά που μας είπε και τη συνεργασία της μαζί με τους Κιώδης. Όντως, ε, πραγματικά η έκθεσή της εστιάζει στα πιο σημαντικά θέματα και νομίζω ε, λόγω και της δημοσιονομικής κρίσης θα πρέπει να περιοριστούμε στα πιο σημαντικά. Έχουμε και την έκθεση του Συμβουλίου στην οποία αναφερθήκατε και νομίζω ότι πολύ δύσκολα ε, θα μπορούσαμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τους ε, κρατικούς ε, προϋπολογισμούς με νέα μέτρα και χρηματοδότηση παρόλο που πρόκειται για επενδύσεις και ανάπτυξη. Είμαι πολύ απογοητευμένος λοιπόν από το Συμβούλιο γιατί έχει άσχημες επιπτώσεις για τις μεταφορές που είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός κλάδος για εμάς. Να σας πω πως ε, βεβαίως όταν δεν συζητάμε το θέμα της ε, χρηματοδότησης μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί, να έχουμε παθές, να συζητάμε με το Συμβούλιο, να καταθέτουμε προτάσεις, προτάσεις σχεδίων, να μιλάμε για την προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία, να μιλάει το Συμβούλιο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τελικά όταν κατευθύνει ο λογαριασμός και πρέπει να τα δούμε όλα στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου προπολογισμού δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα δεν μπορούμε να, κάνουμε, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτές τις ε, γραμμές, αλλά δυστυχώς ε, όλες, όλες έχουν ε, πληγεί με απαράδεκτες, με απαράδεκτες μειώσεις. Ξέρετε πόσοι ήταν οι μείωση στις μεταφορές και στις τηλε, τηλεπικοινωνίες, ήταν εκατομμύρια και Νομίζω ότι όλα αυτά ε, θα πρέπει να τα δούμε υπό την οπτική γωνία και το φως της ανάπτυξης. Έχουμε το προϋπολογισμό για το 2013 και ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν λογική και αυτές οι προτάσεις τροπολογίας νομίζω θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε στις αρχικές και πολύ ρεαλιστικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν φανήκαμε καθόλου μαξιμαλιστές. Ήταν πολύ λογικές οι προτάσεις και ως τελευταίο παράδειγμα θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι μειώσαμε τους προϋπολογισμούς για όλες τις υπηρεσίες. Πώς λοιπόν να έχουμε νέα θαλάσσια πολιτική. Πώς μπορούμε να έχουμε νέες, νέες θαλάσσιες διαδρομές και παρόλα αυτά να μειώνουμε ε, κατά 450 εκατομμύρια τον προπολογισμό μας. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερες ή περισσότερες υπηρεσίες με μειωμένο προπολογισμό. Για τα πειραματικά σχέδια και τα πιλωτικά σχέδια θεωρώ πω οι δύο δράσεις για τον τουρισμό που είχαν προταθεί ε, για μια παράτηση θα πρέπει να διατηρηθούν αλλά δυστυχώς για τον τουρισμό δεν έχουμε συγκεκριμένη πολιτική και πιστεύω πως γνωρίζω γιατί για το e-ticketing δεν διατήρησαν τις προτάσεις γιατί έχουμε μια άλλη προκήρυξη που δεν είναι πιλωτικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ένα project με 9 εκατομμύρια ευρώ, ένα project του e-ticketing. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα κονδύλια αυτά από ό,τι θα ε, είχαμε αν πρόκειται για ένα πειραματικό σχέδιο και δεν μπορούν να τρέξουν και τα δύο ταυτόχρονα, γι' αυτό νομίζω λοιπόν το αφήσαμε στην άκρη. Θα επανέλθουμε, ε, θα έχετε πάρα πολλές τροπολογίες ε, κάθε φορά, όπως έχετε κάθε φορά, αλλά νομίζω ότι ακόμα, φέτος είναι ακόμα πιο σοβαρό γιατί αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα της κρίσης. Κυρία Ρουβιάλη για τους σοσιαλιστές, ευχαριστώ πολύ. Λίγα μπορώ να προσθέσω. Τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και με την κυρία Μέισνερ συναντηθήκαμε για να δούμε ποια θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει η γνωμοδότηση και γενικά συμπεριζόμαστε τις προτάσεις σας. Όντως, η πρόταση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση που έγινε στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι αρκετά απογοητευτική. Είναι μάλλον σαν κακόγουστο αστείο, γιατί έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα που μιλούσαν για την ανάγκη για ένα σύμφωνο ανάπτυξης με 20 δις ευρώ και έχουμε τον προπολογισμό των 150 δις που θα μπορούσαμε να έχουμε και το πρώτο που κάνει το Συμβούλιο είναι να τον περικόπτει και κυρίως στην κατηγορία 1α που έχουμε όλες τις πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα και επίσης στα περιφερειακά ταμεία και στα ταμεία συνοχής. Μήπως θα πρέπει στο Συμβούλιο να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών με τους ε, υπουργούς οικονομικών και τους υπαλλήλους εκεί για το τι ακριβώς θέλουν. Θέλουν να μειώσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή θέλουν να προσθέσουν κονδύλια για την ανάπτυξη. Για τις τροπολογίες, για να επανέλθουμε στις προτάσεις τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η πρόταση αυτή ήταν λογική. Και συμβαδίζει και με τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μία μικρή παράγραφο στη γνωμοδότηση για τις πληρωμές. Γιατί θεωρώ πως αυτά τα 25 εκατομμύρια για το Μάρκο Πόλο ή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που θα περικοπούν δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει δεκτό. Την προηγούμενη φορά είπαμε πως η μεγάλη συζήτηση φέτος θα είναι όχι ανάληψη υποχρεώσεων αλλά οι πιστώσεις πληρωμών. Η Κυπριακή Προεδρία στον τρίλογο του Ιουλίου δεν θα καταφέρει πολλά, θα είναι μια απλή απογραφή των θεσεών μας. Η Προεδρία μόλις έχει αναλάβει τα καθήκοντά της, δεν έχει ακόμα καταλάβει ποια είναι η εντολή ε, από το Συμβούλιο και νομίζω πως ο Επίτροπος Λεβαντός και ήδη μας εξήγησε πως το Σεπτέμβριο θα έχουμε το διορθωτικό προϋπολογισμού με δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε λοιπόν για μικρό ποσά. Εάν πρόκειται λοιπόν να, είμαστε, ε, να έχουμε αυτή την, ε, την ανάγκη να καλύψουμε αυτά τα ε, κάποια δισεκατομμύρια γιατί, είμαστε, γιατί έχουμε κάποιες επιπλέον ανάγκες, πώς μπορούμε να έρθουμε μετά στην συζήτηση εδώ και να πούμε ότι για τον επόμενο προϋπολογισμό θα κάνουμε και άλλες περικοπές. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών γιατί θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω άλλους σκιώδεις. Η κυρία Σανελόβα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω για την έκθεση. Συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε για τον τουρισμό και για τα πειραματικά αυτά σχέδια. Κοιτάξτε, γίνονται περικοπές στον προπολογισμό, ε, ακόμα και για την οδική ασφάλεια και προηγουμένως μας είπαν ότι είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Νομίζω λοιπόν πως αυτό θα πρέπει να απηχείται και από τον προπολογισμό μου και σας ευχαριστώ για το σημείο 6. Θα πρέπει ο προπολογισμό να διατηρηθεί εκεί που ήταν. Ο κ. Τόσμαν την Επιτροπή. Πώς θα γίνει ο τετραγωνισμός του κύκλου ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε και αυτά τα οποία δεν θέλει να δαπανίσει στο Συμβούλιο. Σαφώς δεν θέλει να τα δαπανίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους σας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισήγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περήφανη για αυτό το σχέδιο και για το, το προσχεδίο του προϋπολογισμού. Όπως είπατε, είχαμε μακρότατες συζητήσεις ε, μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής για τον οργανισμό της ε, για την αεροπορία και θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές σε αυτά τα σχέδια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε εξοικονομήσεις και οπότε θέλουμε την πλήρη υποστήριξή σας ε, ε, πάνω σε αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε γιατί έχετε καταγράψει τις προσπάθειες που καταβάλαμε ε, όλοι μας. Ύστερα θέλω να σας πω πάνω σε δύο σημεία τα οποία θέλω να θίξω εδώ για την πιστοποίηση των εργασιών ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έχει, έχει αναλάβει αυτό το σχέδιο από το 2011. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε έτοιμοι το 2013. Ίσως το 2014 θα μπορούμε να, σας, να έχουμε περατώσει μια φάση και να σας μιλήσουμε γι' αυτό. Ίσως χρειαστεί να ε, υπάρξει παράταση. Είναι ένα τεράστιο σχέδιο και τα κονδύλια έχουν διασφαλιστεί τουλάχιστον για ολόκληρο το 2012. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε για την οδική ασφάλεια που είναι μέγιστη προτεραιότητα, δύο λόγια, ίσως να μην είναι ορατό στον προϋπολογισμό αρκετά αυτό. Ξέρετε ότι έχουμε μία γραμμή στο προϋπολογισμό που είναι στην γενική πολιτική μεταφορών μας και για το 2012 αυτή η γραμμή για το έτος 2012 έχει βεβαρηθεί πάρα πολύ, από το, είναι πολύ βεβαρημένη από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, ο οποίο ε, χρειάζεται κονδύλια για το 2013, αλλά μπορούμε να σας διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν ε, πόροι για την οδική ασφάλεια ε, και θα υπάρξουν σε αυτή τη γραμμή που υπάρχει για τις μεταφορές του 2013. Εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Υπόθηκαν όλα. Συμφωνούμε νομίζω ότι η Κομισιόν έκανε καλές προτάσεις. Δεν τα είπα όλα, αλλά φυσικά είναι απαράδεκτο αυτό που είπε το Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι όλοι θέλουν να υπάρξουν οικονομίε, αλλά δεν είναι δυνατόν. Οπότε θα το επιχειρήσουμε να το αποφύγουμε μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ όλου του Σκιώδη, όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ. Θα είναι πρόβλημα γενικότερα και με το Συμβούλιο και με, τις, με το πολιετές πλαίσιο γιατί κοιτάξτε δεν μπορείς να έχει και την πίτα και το σκυλό χορτάτο και δυστυχώς θα μας απαντήσουν πως δεν υπάρχουν τα χρήματα. Λοιπόν, 26 Ιουλίου προθεσμία για τις τροπολογίες 6 Σεπτεμβρίου ψηφίζει η Επιτροπή, Επιτροπή Προπολογισμού 3 με 4 Οκτωβρίου και μετά στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. 26 Ιουλίου λοιπόν, τελική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης και με χαρά σας περιμένω στις 3 σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ.